Euh, euh, euh. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας μάλλον. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Έχουμε την δημόσια κρόση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα ε, της πρόσφατης πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης και της ε, δωροδοκίας ε, και την άμεξη της Όλαφ στις πρωτοβουλίες αυτές. Έχετε λάβει στα αγγλικά το πρόγραμμα. Σήμερα στη συνεδρίασή μας έχουμε διερμηνία από και προς πολλές γλώσσες. Ελπίζω ο καθένας να βρει και το κανάλι που τον ενδιαφέρει. Επίσης, η συνεδρίασή μας αναμεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Παρακαλώ, έχετε υπόψη ότι κάθε φορά που ενεργοποιεί κάποιος το μικρόφωνο, αυτόματα η κάμερα θα στρέφεται προς τον ομιλητή. Ας περάσουμε λοιπόν στην ακροασή μας. Στις 8 Οκτωβρίου, ο αρμόδιος επίτροπος ε, για την Τελωνιακή Ένωση και τη φορολογία, τον έλεγχο και την καταπολέμηση ε, της απάτης, ο Επίτροπος Αλγκύρτας Σεμέτα μας είχε παρουσιάσει τις ε, πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά και μάλιστα την ομιλία του την έχετε λάβει και στο φάκελο με τα σχετικά έγγραφα της σημερινής δημόσιας ακρόασης. Έχουμε τέσσερις καλεσμένους εμπειρογνώμονες σήμερα στη Δημόσια Ακρόαση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρώτο μας προσκεκλημένο, τον κύριο Τζοβάνι Κέσλερ, που είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΟΛΑΦ, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Καταπολέμησης της Απάτης. Κύριε Κέσλερ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ε, ενημερώσω σύντομα και στη συνέχεια να συζητήσουμε μαζί τις ε, πρόσφατες πρωτοβουλίες ε, για της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει το θέμα, αλλά όχι μόνο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα κοινοτικά θεσμικά όργανα συμμετέχουν στην εκπόνηση αυτών των πρωτοβουλειών για την καταπολέμηση της απάτης και της ε, δωροδοκίας. Έχω ένα δεκάλεπτο μόνο στη διάθεσή μου. Έχω μοιράσει την ομιλία μου. Δεν πρόκειται να τη διαβάσω, μια και την έχω δώσει, για να μην σας κουράζω και να μην γίνομαι φορτικός. Θα επιμείνω σε τρία θέματα εν σύντομη και μετά είμαι στη διάθεσή σας ε, για να λύσω τις απορίες και να συζητήσουμε και τα διάφορα θέματα. Τρία είναι τα πιο σημαντικά σημεία αυτή τη στιγμή στο έργο μας είναι η αναθεώρηση του κανονισμού 1073, του κανονισμού δηλαδή για την θέσπιση και τη λειτουργία της ΟΛΑΦ. Φαίνεται ότι ο κανονισμός φτάνει στο πέρας ενός μακροχρόνιου ταξιδιού ο κανονισμός αυτός είναι πολύ σημαντικός, όχι μόνο για την Όλαφ, αλλά και γενικώ για το θέμα της πάταξης, ε, της απάτης, ε, της δωροδοκίας ε, και των ατασταλιών και στα κοινοτικά θεσμικά όργανα, αλλά και στα κράτη-μέλη. Και όχι μόνο στα κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικώ. Επίσης έχουμε την νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μόλις ξεκίνησε την νομοθετική της πορεία, πρόσφατα δηλαδή τον Ιούλιο, για τις ε, ποινικέ κυρώσεις ε, σε περίπτωση απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για μας. Και το τρίτο θέμα είναι η πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, ΕΠΟ, που ξεκίνησε να συζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον επόμενο Ιούνιο θα υποβάλει και την πρόταση κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της απάτης και της ιδωροδοκίας. Τώρα, για τον κανονισμό πρώτα. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερος για τις πρόσφατες αποφάσεις και της δικής σας Επιτροπής. Από ό,τι ξέρω δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η απόφαση. Η οριστική απόφαση φαντάζομαι θα ληφθεί ως νούπο και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και καλό θα ήταν να διαμορφωθεί μια ασφάλεια δικαίου και μια βεβαιότητα και για μας και για τους εταίρους μας το συντομότερο δυνατό δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται, γιατί εσείς είστε οι πρωταγωνιστές ε, του όλου εγχειρήματος, οπότε γνωρίζετε εκ των έσω τα πράγματα. Αυτό που θα μπορούσα να πω από πλευράς Όλαφ είναι ότι ο κανονισμός αυτός ε, με την αναθεώρηση που θα γίνει θα λάβει υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα των ενδιαφερομένων, τη διάρκεια της ε, έρευνας, της ανάκρισης. Τώρα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη δεν υπάρχει ένας πραγματικός μηχανισμός ε, για κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η ειλικρινής μου γνώμη. Βέβαια, με την αναθεώρηση του κανονισμού θα εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για κάποιες διαδικασίες που ήδη ε, εφαρμόζουμε και ακολουθούμε, αλλά με δική μας πρωτοβουλία. Και καλό θα ήταν ε, να υπάρχει και μια νομική βάση για την εφαρμογή τους και στον κανονισμό. Γενικώ ο κανονισμός θα είναι καλός για την Όλαφ, για το έργο μας, για τις έρευνες και την προσπάθεια πάταξης της απάτης. Μην περιμένετε, ούτε κι εγώ το περιμένω. Ας μην προσδοκούμε λοιπόν τίποτα ρηξικέλευτες αλλαγές ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των ερευνών με τον 1023. Το αντίθετο θα έλεγα. Θα έλεγα ότι υπάρχει ήδη μία ορατή και σημαντική αύξηση των ελέγχων του έργου μας. Αυτό το λέω ως, αρνητικό, ως κατερνητικό, είναι θετικό. Υπάρχει αύξηση των εκθέσεων και των αναφορών που καλούμαστε να υποβάλουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Καλό και αυτό. Αλλά αυτό το τμήμα του έργου μας θα αυξηθεί αισθητά. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε πόρους για τη σύνταξη εκθέσεων, για την οργάνωση συσκέψεων, συναντήσεων, ενημερωτικών και το καθεξής. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει κανένα τμήμα του τροποποιημένου κανονισμού που να μας διευκολύνει να, μας, να ενισχύει τις αρμοδιότητές μας στις ε, έρευνες. Αν θέλετε να πούμε κάτι που δεν αφορά το 1023 ιδιαίτερα, αλλά γενικώ τη συζήτηση για τον προπολογισμό, η ΟΛΑΦ, όπως και όλες οι άλλες υπηρεσίες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντιμετωπίζει περικοπές ε, της τάξης του 2% κάθε χρόνο για μια πενταετία. Οπότε θα συρρυκνωθούν οι πόροι μας, ενώ ταυτόχρονα θα συρρυκνωθούν και οι ανθρώπινοι πόροι και με το 1073 θα χρειαστεί να αφιερώσουμε περισσότερους υπαλλήλου μας στη σύνταξη εκθέσεων. Οπότε θα χαθεί προσωπικό από τις έρευνες. Άρα θα γίνουν πιο αναποτελεσματικές. Παρόλο που συγκεντρώνουμε τις έρευνές μας, αλλά και κάποιοι κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ότι πριν κλείσουμε την έρευνα θα πρέπει να έχουμε ακρόαση ενδιαφερομένου. Και τι γίνεται σε περίπτωση που εκκρεμωδικεί αλλού η υπόθεση. Αυτό μας εμποδίζει και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να, περιμένουμε. Αυτό θα καταστεί ακόμη πιο χρονοβόρα τη δική μας έρευνα. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Φέτος θα έχουμε 30% περισσότερες πληροφορίες ή καταγγελίες για δωροδοκίες και απάτες. Πέρυσι είχαμε 1046 καταγγελίες και μάλιστα πολλές από αυτές ε, είναι αβάσιμες, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όλες αυτές τις 1046 ε, καταγγελίες να τις διαλευκάνουμε. Και μάλιστα φτάσαμε σε ένα ρεκόρ της ΟΛΑΦ σε ό,τι αφορά τη σειρόη. Φέτος έχουμε πάνω από χίλιες πάλι καταγγελίες και κάναμε έναν απλό μαθηματικό υπολογισμό που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε πάνω από 1.300 συνολικά καταγγελίες. Δεν μπορούμε να τις αρχιοθετήσουμε, θα πρέπει όλες να τις αναλύσουμε και να εξακριβώσουμε κατά πόσο ευσταθούν. Οπότε έχουμε αυξημένο έργο, λιγότερο προσωπικό και έχουμε δαπάνες ενό εκατομμυρίου και για διοικητικά έξοδα, αλλά δεν, δεν είναι δυνάμεθα να το χρησιμοποιήσουμε για το προσωπικό. Οπότε με το 1073 έχουμε περισσότερε υποχρεώσει, αυξημένε υποχρεώσει διοικητικέ και υποβολή εκθέσεων και, λιγότερο προσωπικό. Οπότε θα έκανα μια πρόβλεψη για τις ερευνητικές δυνατότητες της ΟΛΑΦ για το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι μάλλον αρνητικές αυτές οι προβλέψεις. Πάντως, καλό είναι που με την αναθεώρηση του κανονισμού 1073 θα έχουμε ένα νέο πλαίσιο και θα εγκριθεί τελικά η αναθεώρηση αυτή, αλλά ίσως θα πρέπει να ληφθούν και συμπληρωματικά μέτρα, τουλάχιστον να μην ε, ε, περιοριστεί το προσωπικό. Μη μου κόβετε προσωπικό. Δεν λέω ότι το κόβετε εσείς προσωπικά, αλλά τουλάχιστον να μπορέσω να χρησιμοποιήσω τις οικονομίες μας από τι διοικητικέ δαπάνε για να κρατήσουμε τους υπαλλήλους που έχουμε τώρα. Να μην περικοπεί ακόμη το προσωπικό μας. Αυτά ως προς τις αλλαγές του 1073 και τον αντίκτυπο που θα έχει η τροπολογία του κανονισμού στις ερευνητικές ικανότητες ε, της ΟΛΑΦ. Δεύτερο θέμα Ήδη σα ενημέρωσε για το δεύτερο αυτό θέμα την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε την νομοθετική πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που την εκπώνησαν οι ΟΛΑΦ από κοινού με την Γενική Διεύθυνση Just Δικαιοσύνη για την εναρμόνιση της, για την πρόταση της οδηγίας ε, με θέμα την εναρμόνιση του ουσιαστικού ποινικού δικαίου των κρατών μελών για θέματα δωροδοκίας και απάτης, διαφθοράς και απάτης, ε, εφόσον πρόκειται για, οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν μπορούμε ακόμη να έχουμε κάποια φαινόμενα που είναι αξιόπινα σε ορισμένες χώρες και όχι σε άλλες. Υπάρχουν ακόμη τεράστιες διαφορές ε, στις ποινικέ διατάξεις των κρατών μελών, γιατί το αντικείμενο είναι το ίδιο. Είναι κοινοτικά κονδύλια είναι τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κοινό το συμφέρον και άρα θα πρέπει να έχουμε κοινή αντίδραση, κοινή υπεράσπιση, κοινή προσ... προσπάθεια και προστασία και κοινή μέρημνα. Δεν έχουμε λοιπόν μόνο μία μέρημνα, μία εναρμόνιση για μία συμπεριφορά που κρίνεται αξιόπινη σε όλες τις χώρες, γιατί μία σύγκρουση συμφερόντων για τις δημόσιες προμήθειες, για παράδειγμα, δεν είναι έγκλημα σε όλες τις χώρες, αλλά υπάρχει μια ενορμόνιση κάποιων ποινικών διατάξεων. Επίσης, ως προς τις κυρώσεις, μερικές φορές οι παραβάτες εκμεταλλεύονται τις διαφορές στο ποινικό δίκαιο των χωρών μελών. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται και ε, κάποια θέματα προθεσμιών, που συστηματικά εκμεταλλεύονται οι παραβάτες, οι εγκληματίες που συστικά επιλέγουν την δικαιοδοσία, την ομοθεσία, κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αυτό το, το δίνεται να το πράξουν οι εγκληματίες και το κάνουν. Εκμεταλλεύονται την ε, επικέστερη νομοθεσία. Εμείς θεωρούμε τέτοια παραθυράκια είναι απαράδεκτα και με το νομικό εργαλείο της οδηγίας ε, πιστεύουμε ότι θα εξασφαλιστεί μια εναρμόνιση. Υπάρχουν και τα θέματα των ελάχιστων ε, ποινών, ή των ελάχιστων κυρώσεων. Είναι μια έννοια που μερικές φορές ε, δεν υπάρχει στα κράτη-μέλη. Αλλά δεν είναι τόσο κακό όσο ακούγεται. Μπορούμε πολύ εύκολα να εξηγήσουμε και να συμπεριλάβουμε και αυτό το θέμα των ελάχιστων ποινών ή των ελάχιστων ποινικών κυρώσεων. Ελπίζω θα έχουμε την ευκαιρία και στο Κοινοβούλιο να το κάνουμε, να εξηγήσουμε την αναγκαιότητα και αυτή τη διάταξη. Και τρίτο θέμα, το θέμα τη Ευρωπαϊκή Αγγελική Αρχή. ΕΠΟ. Ξέρετε ότι η ίδια συνθήκη κατοχυρώνει ε, με μια διάταξη αυτή την ε, Ευρωπαϊκή Αγγελική Αρχή και οι Επίτροπη Σέμετα και Ρέντινγκ είπαν ότι μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει σχετική πρόταση. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει τη μορφή του κανονισμού. Η ΟΛΑΦ και η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης είναι συναρμόδιες για το θέμα αυτό και συνεργαζόμαστε σε προκαταρκτικό στάδιο, έλεγχο, έλεγχο αντικτύπου, μελέτη επιπτώσεων. Γίνεται ήδη μια προεργασία με συνεργασία ΟΛΑΦ και Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης. Δεν μπορώ τώρα να σας αναλύσω τις λεπτομέρειες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ευελπιστώ ότι σχετικά σύντομα θα μου πείτε και εσείς πότε σκοπεύετε η δική σας επιτροπή μια άλλη επιτροπή, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει επιμερισμένη αρμοδιότητα επιτροπών εδώ για το θέμα αυτό. Να μου πείτε λοιπόν αν θεωρείτε σκόπιμο, ακόμη και σε αυτή την προκαταρκτική φάση, να έχουμε κάποια ανταλλαγή απόψεων, κάποια συνεννόηση, για να δούμε ποιες είναι οι απόψει μα και οι προσεγγίσει μα. Αυτό κάνουμε και στα κράτη-μέλη. Έχουμε κάποιε προκαταρκτικέ συναντήσει με την κυρία Λεμπάκη, τη Γενική Διευθύντρια τη ε, Διάθεση Just. Έχουμε πάει και μαζί και ξεχωριστά σε διάφορε πρωτεύουσε. Και αυτή τη βδομάδα επίση έχουμε επισκέψει δύο πρωτεύουσε. Πρόκειται για μια άτυπη προκαταρκτική ανταλλαγή απόψεων. Και φυσικά και το Κοινοβούλιο και τα κρατημέλη θα έχουν την ε, δυνατότητα επίσημα να σχολιάσουν την πρόταση μετά την επίσημη υποβολή της τον Ιούνιο. Εμείς όμως κρίναμε σκόπιμο και σε αυτή την προκαταρκτική φάση να ξεκινήσουμε μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων και με τα κράτη-μέλη και βελτιστούμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί θεωρώ ότι αυτή είναι μια απαραίτητη λύση που θα αντιμετωπίσει και πάλι το πρόβλημα της συνεργασίας ε, των ε, κρατών με την ΟΛΑΦ, το θέμα της αποτελεσματικότητας των ερευνών. Με τον κανονισμό δεν θα μπορούσαμε να έχουμε άλλες αλλαγές. Εμείς ε, χορηγούμε τις ερευνές μας στα πορίσματά μας σε εθνικές αρχές, στους ε, εισαγγελείς, στα κράτη-μέλη και εκείνοι από ε, άποψη ποινικού δικαίου θα πρέπει να ξαναρχίσει τη διαδικασία και την ανάκριση από την αρχή. Και μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο πρόθυμοι, περισσότερο ή λιγότερο ικανοί να την φέρουν σε πέρας και στην καλύτερη περίπτωση χάνουμε αμήντε άλλο χρόνο. Δεν παραπονιέμαι, απλώς σας παρουσιάζω την κατάσταση. Εμείς κάνουμε κάποιες διοικητικές ε, έρευνες. Εμείς δεν έχουμε πρόσβαση ε, σε πληροφορίες ενός τραπεζικού λογαριασμού, για παράδειγμα. Οπότε πώς μπορώ να ερευνήσω εγώ για απάτη ή για διαφθορά αν δεν έχω πρόσβαση σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Εν πάση αυτό σας το λέω ενημερωτικά. Προσπαθούμε να έχουμε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Οπότε, σε περίπτωση που θεσπιστεί αυτό το Ευρωπαϊκό Γραφείο ε, εισαγγελία, θα παρακάμψουμε τέτοιες δυσκολίες. Και αυτό δεν θα σημαίνει έλλειψη από απώλεια κυριαρχίας από τα κράτη-μέλη. Παρακαλώ να μην παρεξηγηθούμε. Ένα από τα μοντέλα που εξετάζουμε και βλέπουμε ότι τη χάνει τις μεγαλύτερες υποδοχές και στα κράτη-μέλη είναι το γραφείο αυτό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα να απαρτίζεται από ένα κεντρικό γραφείο και από, από, εισαγγελείς, από εθνικούς εισαγγελείς. Θα είναι ουσιαστικά δηλαδή ένα δίκτυο εθνικών ε, εισαγγελικών γραφείων με το πανευρωπαϊκό με συνεργασία. Και γιατί χρειαζόμαστε μια τέτοια Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή πέραν των προβλημάτων της ΟΛΑΦ και των ερευνών. Όπως είχα την ευκαιρία να σας πω και σε άλλη περίπτωση στην Επιτροπή Κρίμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέτοιου είδους ε, εγκλήματα, απάτες, διαφθορά, δωροδοκία, πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκφύσεως έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Ε, πρόκειται για πανευρωπαϊκά ουσιαστικά εγκλήματα και αν συνεχίσουμε, όπως τώρα δηλαδή, να τα αντιμετωπίζουμε με εθνική μονοπροσέγγιση, με εθνικά μέσα, με εθνικούς φορείς και όργανα, όπως κάναμε από τον 19ο αιώνα και έχουν περάσει δύο αιώνες και το ίδιο πράγμα κάνουμε. Με τις ε, ερευνητικές επιτροπές, τον ανακριτή. Βέβαια, έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση, αλλά ελάχιστα. Είναι σαν να κανείς ένα παλαιό αυτοκίνητο που έχει, το αγαπάει ιδιαίτερα γιατί έχει συναισθηματική, ε, συναισθηματικό δεσμό μαζί του. Μπορεί να το περιποιείται και να το βελτιώνει, αλλά εξακολουθεί να είναι το παλιό αυτοκίνητο. Το ίδιο κάνουμε. Συνεχίζουμε δηλαδή να αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που έχει αλλάξει ριζικά και έχει ξεπεράσει τον εθνικό της χαρακτήρα, έχει αποκτήσει ένα διασυνοριακό χαρακτήρα, γιατί αυτό το χαρακτήρα έχουν τα οικονομικά εγκλήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τα αντιμετωπίζουμε με εθνικό τρόπο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Απλή απάτη, έρευνα της ΟΛΑΦ. Μια ε, υπόθεση που έφτασε και στις εφημερίδες, μπορώ να σας ενημερώσω. Και το είχα πει και στην επιτροπή σας σε μια ακρόαση που είχατε για μια γερμανική περίπτωση. Έρευνα της ΟΛΑΦ. Απλή περίπτωση απάτης, εκατομμυρίων βέβαια, ε, για υπερτιμημένα τιμολόγια που ε, χρησιμοποιούσαν βούλγαροι επιχειρηματίες. Εμείς ανακαλύψαμε την απάτη. Ποιος όμως ε, συνέτασε τα τιμολόγια. Ένας Γερμανός επιχειρηματίας, γερμανική επιχείρηση. Με το σύστημα του 19ου αιώνα λοιπόν που χρησιμοποιούμε το στείλαμε σε δύο εισαγγελίε. Στη γερμανική για το γερμανικό τμήμα, στη βουλγαρική εισαγγελική αρχή για το βουλγαρικό τμήμα. Εθνικό, εθνική προσέγγιση, δύο χώρε. Βέβαια, τα τεκμήρια, οι αποδείξεις, τα αποδεικτικά στοιχεία είναι τα ίδια. Το έγκλημα είναι το ίδιο. Ένα έγκλημα που διέπραξαν από κοινού δύο ε, αυτούργοι. Δύο όμως ε, ανακρίσεις, δύο δίκες είναι μη τι άλλο χρονοβόρα διαδικασία. Και στην περίπτωση αυτή είχαμε και δύο διαφορετικά αποτελέσματα. Ήταν δίκαιο, αυτό, δύο διαφορετικέ εκβάσει. Όχι, κάποιο έκανε λάθο. Αλλά τέτοιου είδου αποτελέσματα τα βλέπουμε, για να μην πω καθημερινά, κάθε ένα-δύο μήνε. Πολύ συχνά πάντω. Σε μερικέ περιπτώσει έχουμε διαφθορά που διαπράτεται σε μία χώρα, αλλά ε, τα χρήματα έχουν πληρωθεί σε μια τρίτη χώρα ή από μια τρίτη σε τέταρτη και έχουν καταλήξει σε μια πέμπτη χώρα σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Σε μια χώρα όμως που η νομοποίηση παράνομων εσόδων δεν θεωρείται αξιόπινη πράξη. Οπότε ποια είναι η αρμόδια δικαιοδοσία και ποια είναι η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ποιος μπορεί να δει το έγκλημα. Εμείς επειδή έχουμε την ευρωπαϊκή προοπτική, το βλέπουμε. Αλλά σε εθνικό επίπεδο βλέπουν μόνο μια κίνηση κονδυλίων, χρημάτων, κεφαλών και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Αν κανείς περιορίζεται στο στενό εθνικό πρίσμα, δεν μπορεί να δει την όλη κατάσταση. Εμείς την αντιληφθήκαμε, γιατί έχουμε αυτή την πανευρωπαϊκή προσέγγιση, αλλά διαπιστώσαμε ότι δεν είχαμε τη δικαιοδοσία. Κάθε χώρα περιορίζεται στη δική της ε, εθνική επικράτεια σταματάει στα σύνορα η δικαιοδοσία της. Οπότε ουσιαστικά είχαμε μια αρνητική ε, σύγκρουση δικαιοδοσιών ή συγκρόμενες δικαιοδοσίες ή αντικρουόμενα αποτελέσματα δικαιοδοσίας. Η απάντηση σε όλα αυτά τα προβλήματα είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Προφανέστατη απάντηση και μάλιστα επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί το συντομότερο δυνατό αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Γιατί το ίδιο ισχύει και για το λαθρεμπόριο. Και αυτό εξορισμού έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Και, και οι Λιθουανοί που υποφέρουν γιατί έχουν εκτεθειμένα σύνορα και με την Πολωνία πρέπει να το αντιμετωπίσουν, αλλά έχουν τέσσερις εισαγγελικές αρχές. Γιατί ό,τι μπαίνει από τη Λιθουανία και την Πολωνία κατευθύνεται προς τη Γερμανία ή σε άλλες πέντε χώρες, οπότε θα πρέπει να επιμερίσουν την έρευνα και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουν κάτι που εξορισμού ορισμού εκφύσεως έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί κάτι διασυνοριακό με κατακαιρματισμένο εθνικό τρόπο. Μια Ευρωπαϊκή λοιπόν εισαγγελική αρχή, ένα ε, γραφείο του Ευρωπαίου εισαγγελέα θα αποτελέσει την απάντηση γιατί είναι διασυνοριακά τα εγκλήματα, είναι κοινά τα συμφέροντα, είναι τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε χρήζουν και κοινή απάντηση. Ελπίζω να με ακρηγόρησα, είμαι στη διάθεσή σας για να λύσω κάποιες απορίες ή να έχουμε συζήτηση και ελπίζω είτε με τη δική σας επιτροπή είτε οπουδήποτε αλλού να συζητήσουμε πιο εμπεριστατωμένα το θέμα του ΕΠΟ, της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζοβάνι Κέσλερ. Πάμε αμέσω στην κυρία Γιάννα Μαγερ, επικεφαλής του Βελγικού Γραφείου του Transparency International, που θα εκφράσει μια άποψη εκ των έξω, την εξωτερική πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. για το θέμα. Je vous invite euh, alla tribuna. Oui, alors, euh, Κύριε Γιάννα Μίτερμαϊ, λοιπόν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Ευχαριστώ που καλέσατε την Transparency International να μιλήσει επ' αυτή την ευκαιρία. Καλώς ορίζω αυτή την ευκαιρία να εκφράσω μια άποψη εκ των έξω. Από πλευρά κοινωνία των πολιτών για αυτά τα σημαντικότατα θέματα, σημαντικότατες μεταρρυθμίσεις που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα εκτιμούμε τι πρωτοβουλίε δηλαδή υπάρχει νέα πρόταση για την καταπολέμηση της απάτης μέσω του ποινικού δικαίου. Αυτό το θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό βήμα. Και δεύτερον, το επόμενο έτος, τον Ιούνιο, θα ξεκινήσει η έκθεση καταπολέμησης διαφθοράς ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταπολέμηση διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί ασχολείται με τις ε, κρατικές και αυτό σχετίζεται άμεσα με την χρήση των ευρωπαϊκών πόρων σε εθνικό επίπεδο και κάποιοι πολιτικοί πράγματι έχουν πρόθεση ε, να προωθήσουν τη δημιουργία του, της Αγγελικού Γραφείου, του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα και επίσης και το θέμα της κατάσχεσης ε, των προϊόντων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετικές και έτσι διαφυλάσσονται οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από την διαφθορά και από την απάτη που, ποια ζητήματα τίθενται σε σχέση με αυτά που προανέφερα. Ε, βλέπουμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και θεωρούμε ότι οι σε αυτές πρωτοβουλίες, οι προταθήσεις πρωτοβουλίες θέτουν ένα ανομικό πλαίσιο εξετάζουν τα θέματα δίωξη ε, κύρωση. Ε, ε, ανάκτησης παρανόμων εσόδων και το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να υπάρχει όσον αφορά τη διαφάνεια, ε, ε υποβολή αναφοράων, ε, έρευνες κλπ. όπως ανέφερε και Όλεφ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, διότι οι πρωτοβουλίες λαμβάνουν υπόψη κάποιες στοιχές μόνο, όχι όλες, και υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη για περισσότερες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να προστατευτούν οι πόλεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, πλήρως. Ας μπούμε τι παραπάνω μπορεί να γίνει. Ας προχωρήσουμε καταρχάς στο θέμα της διαφάνειας. Πολλές με κυβερνητικές οργανώσεις, όχι μόνο η Transparency International, επανειλημμένα ζήτησαν μία ε, ενιαία, ένα πλήρες σύστημα ενιαίο στο διαδίκτυο online, όπου ε, να δημοσιεύονται όσοι πληροφορίες, όχι με κατακαιρματισμένο τρόπο, να δίνονται πληροφορίες επί διαφόρων, για διάφορε σελίδε που ε, προωθούν τα διάφορα κατημέλια αλλά σε μια ιστοσελίδα να διατίθεται πληροφορίε. Και δεν χρειάζεται κατακαιρματισμός των πληροφοριών. Θέλουμε ενιαία απειλή, μια ιστοσελίδα θα δείχνει τον προπολογισμό, τα κονδύλια, σαφείς ενδείξεις των πόρων που θα δαπανηθούν και προς πού πηγαίνουν, κατευθύνονται τα χρήματα. Όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική ή τα διεθνωτικά ταμεία για την επόμενη περίοδο, Δεν προβλέπεται τίποτα για μια κεντρική βάση δεδομένων για αυτά τα ταμεία, για αυτούς τους πόρους. Ούτε για τους τομείς, ούτε για το σύστημα στο σύνολό τους. Οπότε, σαν οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, ανησυχούμε ότι αυτή η κατακαιρματισμένη χρηματοδότηση δεν διευκολύνει τον έλεγχο χρήσεως των πόρων και τελικά ε, η εικόνα σχετικά με τι ροέ των χρημάτων ε, παραμένει θολή και υπάρχει κάποιο κενό όσον αφορά την προστασία των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν μπορούμε μόνο να επικρίνουμε τα χρήματα το πώς δαπανώνται, 80% των χρημάτων που δαπανώνται από τα κράτη-μέλη, στα πλαίσια της κοινής διαχείρισης, ε, βλέπουμε και ποια χρήματα δαπανώνται άμεσα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ οι συνάδελφοι έχουν δημοσιεύσει έναν ενδεικτικό κατάλογο των δαπανών και ποια χρήματα πηγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρε χώρες και πώς γίνεται διαφανής χειρισμός αυτών. Βρήκαμε ότι υπάρχουν κενά όσον αφορά τη διαφάνεια των πόρων που δίνουν στις χώρες της διεύρυνσης, υποψηφίων και ενδεχομένω υποψηφίων χωρών. Όσον αφορά τα χρήματα που πηγαίνουν εκεί, βλέπουμε ότι όσον αφορά τη διαφάνεια επιδόσει είναι κακές και χρειάζονται κατεπηγόντως κάποιες κινήσεις, κάποιες δράσεις για να καλυφθεί το κενό για να συνοψίσω για τα προβλήματα που έχουμε όσον αφορά τη διαφάνεια, αυτό που χρειάζεται, για να το επαναλάβω σαφώς και να το πω δυνατά για να το ακούσετε όλο, ενιαία στο σελίδα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, όπου φαίνονται όλοι οι δικαιούχοι που δέχονται του πόρου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και δημοσιεύονται. Ήρθα στι Βρυξέλλε πριν από 4,5 χρόνια ε, και ήταν από τι πρώτε συστάσει που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έγινε κάτι γι' αυτό. Τέλο πάντων, Κάποια κράτη-μέλη βέβαια αύξησαν τη διαφάνεια όσον αφορά τους δικούς τους δικαιούχους, αλλά τίποτα δεν άλλαξε όσον αφορά τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος. Και τώρα ερχόμαστε στη δεύτερη δυναμία που λείπει από τις πρωτοβουλίες και αφορά την υποβολή αναφορών. Ε, είναι ένα θέμα ε, το οποίο το έχει παρατηρήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια. Θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το τομέα διότι το σύστημα επικοινωνία των κρατών μελών και υποβολή αναφορών από κάτω μέσα σε κράτο μέλος ποικίλει και οι διάφορε υποθέσεις που αναφέρθηκαν από τα κράτη-μέλη και αναφέρθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ λίγες. Ένας λόγος γι' αυτό, σύμφωνα με την αξιολόγησή μας, είναι γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλοι διευλοί για την υποβολή αναφορών, απατών, διαφθορά όσον αφορά την χρήση των πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση διότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί υποβολής αναφορών και ενημέρωση ε, με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την κοινωνία των πολιτών. Δεν συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία κοινωνία των πολιτών. Η Transparency International έχει ένα κέντρο πολιτών όπου μπορούν να έρθουν και να κάνουν καταγγελίες οι πολίτες όσον αφορά περιπτώσεις διαφθοράς που έχουν διαπιστώσει και δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κέντρου μας, του ε, ΙΛΕΞ και, του, και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό μπορεί να ε, βελτιωθεί και, και άλλες μη κοινωνικές οργανώσεις έχουν ανάλογες ε, πρωτοβουλίες και οι καταγγελίες, πώς καταγγέλλονται αυτές οι τασταλίες είναι ένα πρόβλημα και όσον αφορά τι ε, κρατικέ προμήθειε, υπάρχει νέα οδηγία, η οποία συζητείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία των πληροφοριοδοτών θα μπορούσε να συμπεριληφθεί. Α δούμε τι θα συμβεί του επόμενου μήνε όταν θα υιοθετηθούν αυτέ ε, οι οδηγίε από τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι άλλο όσον αφορά την ενημάζωση πληροφορία ε, και καταγγελίε είναι η σχέση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων με την Όλαφ. Ο, ο κύριο Κέσλερ συνόψισε τις μεταρρυθμίσεις της Όλαφ και τι συνέπειες επιφέρουν αυτές οι αλλαγές, εμείς θα λέγαμε ότι ένα από τα θετικά της μεταρρύθμισης της Όλαφ είναι ότι τουλάχιστον προβλέπεται ότι η σχέση μεταξύ κρατών μελών και Όλαφ πρέπει να ενισχυθεί. Τώρα αν αυτό θα συμβεί στην πράξη είτε όχι είμαι περίεργη, περιμένω να δω σε μερικούς μήνες ή χρόνια. Αλλά αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα συστήναμε και το Συμβούλιο έχει προτείνει, όπως βλέπετε και στην διαφάνειά μας. Για να συνοψίσω λοιπόν, χρειαζόμαστε προστασία των πληροφοριωτών, χρειαζόμαστε ε, κρατικές ε, ε, προμήθειες που θα αντικατοπτρίζουν αυτή η προσπάθεια που γίνεται και θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών στη διαδικασία αυτή και να μην παραμείνει μόνο σε θεσμικό επίπεδο η προστασία των πόρων της Ένωσης. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι η δίωξη και οι έρευνες και αυτό δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στις παρούσες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα θέλαμε να δούμε όπως και όλα να δημιουργηθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ε, αυτό είναι κάτι που εκκρεμεί επί πολλά χρόνια. Δεν υπήρξε επαρκή πολιτική προθυμία ούτε ώστε να υλοποιηθεί η δημιουργία αυτή τη ε, υπηρεσία. Αλλά συμφωνούμε με την αξιολόγηση τη Όλαφ ότι οι διασυνοριακέ περιπτώσει διαφθορά και απάτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επηρεάζουν, που πλήττουν τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα πρέπει να ε, βελτιωθεί η συνεργασία η διακρατική και η διαπεριφερειακή και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να συμβεί. Ανησυχούμε και για αυτό που είπε ο κύριος Κέσλερ ότι μεγαλύτερο ο φόρτο εργασία ε, που περιμένει την Όλαφ και μειώνεται το προσωπικό και το δυναμικό, αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αν αυτό είναι μία από τις συνέπειε μεταρρύθμισης τη Όλαφ, πρέπει να επαναξεταστεί η μεταρρύθμιση της, πιστεύω. Σε έναν κόσμο που περιφερειοποιείται και παγκοσμιοποιείται όλο και περισσότερο. Ε, χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εισαγγελία. Χρειαζόμαστε και πίεση από των κρατών μελών για να εφαρμοστούν όλε οι μεταρρυθμίσει, διότι αν έχουμε πολλού νέου κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και δεν εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη, τι θα συμβεί. Και τέλο, ε, απευθύνω έκκληση να συμπεριθούν οι πολίτε κυρίως και οι ερευνητές δημοσιογράφοι σε, αυτά τα, σε αυτές τις έρευνες να δημιουργηθούν δυνατότητες για αυτούς να εργαστούν, να συνεργαστούν για να βελτιωθεί ο έλεγχος, η διαφάνεια, η υποβολή αναφορών ε, και να καταπολεμηθεί καλύτερη απάτη και διαφθορά στο μέλλον. Απάτη και διαφθορά μπορεί να πλήξουν τους πόρους Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Μίτερμαϊερ. Θα δώσω το λόγο στον το πρόσωπο που ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ακρόαση, τον κύριο Γένς Γκάιερ, μετά από πρωτοβουλία δική του, το των σοσιαλδημοκρατών δηλαδή, έχουμε σήμερα, διεξάγουμε σήμερα την ακρόαση αυτή. Δεν μπορούσα να σας δώσω το λόγο πρώτον, πρώτο πρώτο δηλαδή, αλλά τώρα λαμβάνει το λόγο κύριο Γένς Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προτιμούσα βέβαια να μην είχατε δώσει τον λόγο στην αρχή, πριν από την έναρξη της ακροάσεως. Σίγουρα θα είχατε κάποιους σημαντικούς λόγους που δεν το πράξατε. Ε, θα μπορούσα βέβαια εγώ, αν μου είχατε δώσει τον λόγο στην αρχή, να οργανώσω λίγο καλύτερα τη συζήτηση. Τώρα βεβαίως θα συνεχίσει όπως συνεχίζεται, θα έχουμε ερωτήσεις προς τους δύο πρώτους προσκεκλημένους ειδήμονες. Κύριε Κέσλερ, αντελήφθη ότι μας είπατε ευγενικά μεν, καθαρά δε, ότι ένας από τους στόχους μας, δηλαδή το περισσότερο προσωπικό για τις έρευνες, ότι τον υπονομεύουμε, ζητώντας από εσά περισσότερες εκθέσεις αναφορές ή πάντως επιβάλλοντα περισσότερες απαιτήσει στην Όλαφ που ίσως σας, ε, επιβάλλουν υπερβολικό φόρτο εργασίας. Από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα της πολιτικής αποτελεσματικότητας της εργασίας της Όλαφ. Διότι βεβαίως εμείς τα πράγματα αυτά δεν τα κάνουμε επειδή βαριόμαστε και δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε. Τα ζητούμε αυτά γιατί θέλουμε η αποτελεσματικότητα των ερευνών της Όλαφ να αυξηθεί και μάλιστα με τρόπο διαρκή. Επίσης αντελήφθην ότι αναμένεται πολλά από την ενοποιημένη αυτή Ευρωπαϊκή Διοκτική Αρχή, η Εισαγγελική Αρχή. Αυτό και εμείς το κάνουμε και εμείς αναμένουμε πολλά Θέλουμε όμως από εσά να μάθουμε ποια είναι τα προβλήματα εκείνα που πρέπει να επιληθούν και ποιες είναι οι καλύτερες λύσεις κατά τη γνώμη σας. Αναφέρατε χτυπητά παραδείγματα για περιπτώσεις όπου τουλάχιστον το αρνητικό είναι ότι χάνεται πολύς χρόνος, όταν δηλαδή επεξεργάζονται κάθε ένα μέρος της διώξεως μία χώρα μέλος ξεχωριστά, ή καμιά φορά μάλιστα πάβει η δίωξη. Οι εισαγγελίε των χωρών μελών καμιά φορά αδιαφορούν. Αυτό είναι που εμένα με απασχολεί σε όλη αυτή την ακρόαση. Αν μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα ποιες αρμοδιότητες, ποιες δικαιοδοσίες θα πρέπει να διαθέτει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Τότε καθήκον του Κοινοβουλίου θα είναι βεβαίως να τις εξασφαλίσει αυτές. Αναφέρατε το παράδειγμα της πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά ίσως δεν είναι το μοναδικό. Γι' αυτό να μας πείτε, εφόσον μπορείτε, πιο συγκεκριμένα για το τι θα πρέπει να μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Αυτά για μας θα είναι βέβαια σημαντικότατες υποδείξεις για την παραπέρα εργασία μας. Για την κυρία Μίτα Μάιερ τώρα, την υπόδειξή σας για την κοινή ιστοσελίδα την σημειώνουμε. Και εμείς δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι με την κατάσταση αυτή, δηλαδή με τον κατακαιρματισμό αυτό των, ε, της παροχής πληροφοριών από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όταν μάλιστα κάποιοι δικαιούχοι έχουν λάβει χρήματα ευρωπαϊκά, όπως για παράδειγμα στο Interreg, από διάφορες χώρες, δικαιούχοι από διάφορε χώρε, τότε βεβαίω είναι πάρα πολύ δυσδιάκριτα τα πράγματα. Σημείωσα βέβαια και την ανάγκη συνεργασίας με τις χώρες μέλη που αναφέρατε. Εάν τώρα μπορείτε να, μας, να μου απαντήσετε την ίδια ερώτηση την οποία πήφθηνα στον κύριο Κέσλερ, δηλαδή τι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή να μπορεί να κάνει, τι θα πρέπει να μπορεί να κάνει, ποιες αρμοδιότητες θα πρέπει να διαθέτει για να μπορεί να διώξει ε, υποθέσεις διασυνοριακής απάτης. Πιστεύω ότι εσείς μπορείτε να ε, μιλήσετε πιο ελεύθερα από ότι ο Γενικός Διευθυντής της ε, Όλαφ που είναι αξιωματούχος θεσμικού οργάνου. Γι' αυτό αναμένω από εσά να μου πείτε πιο καθαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Γκέιερ. Θα ήθελα να σας πω ότι από τεχνικό λάθος ε, δεν σας έδωσα πρώτο το λόγο. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν έγινε και εμένα. Δεν είχα καμία πρόθεση να σας παραλείψω. Ας γίνει συζήτηση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμένα η ιδέα του κυρίου Γκάιερ μου φάνηκε εξαιρετικά καλή, διότι η Κομισιόν πριν από τις θερινές διακοπές είχε υποβάλει το σχέδιο αυτού κανονισμού που εμένα μου φαίνεται ρηξικέλευτο πραγματικά. Δηλαδή αποσκοπεί στην βελτίωση μιας καταστάσεως την οποία εφιστάμεθα εδώ και δεκάδες χρόνια, εδώ και δεκαετίες και είναι ανυπόφορη, διότι λαμβάνουμε γνώση για υποθέσεις όπου περιέχονται αξιόπινες πράξεις και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Νομίζω λοιπόν ότι πρόκειται για ορόσημο. Είναι πραγματικά εξαιρετική η πρόταση αυτή. Και γι' αυτό χρειάζεται τώρα να προωθηθεί και βλέπω ότι γίνεται ήδη η προσπάθεια από ορισμένε χώρες ώστε να μην προχωρήσει. Κυρίε και κύριοι, δεν είμαστε αρκετά αυστηροί, διότι θα μπορούσαμε να πούμε όποιος δεν διαχειρίζεται έντιμα τα χρήματα της Ένωσης δεν θα ξαναπάρει άλλα. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε. Και είμαι βεβαία τότε ότι οι χώρες μέλη θα δράσουν ταχύτατα για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Για πρώτη φορά το 2011 έχουμε αριθμούς για το τι κάνει η Όλαφ με τις υποθέσεις που σημαίνουν διάφορες χώρες μέλη. Έχουμε για τη Μάλτα 0% μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Το ίδιο ισχύει για την Λιθουανία, Κύπρο, αν και υπήρξε μία υπόθεση, Σλοβενία 2, άλλες βλέπω 10% Ουγγαρία επίσης πολύ χαμηλό επίπεδο ή κάτω από 14% στη Βουλγαρία 20% στην ε, Πολωνία 22% στην Πορτογαλία ε, εγώ νομίζω ότι και πάνω από 5% θα έπρεπε να είναι ο μέσος όρος είναι 46% των υποθέσεων αυτών στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση κύριε Γενική Διευθυντά εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας ότι με τον νέο κανονισμό της Όλαφ σε αυτόν περιλαμβάνονται πράγματα που δεν θα αποδώσουν τίποτα. Αυτή η ετήσια συνάντηση με το Συμβούλιο για την αντιμετώπιση των απατών θα δείτε ότι αποτελεί και θα αποτελέσει πολύ μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Εσείς είστε σχετικά νέος και γι' αυτό επιτρέψτε μου, όποιος μας γνωρίζει και όποιος γνωρίζει και το Συμβούλιο και όποιος γνωρίζει πώς εμείς διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο, θα γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν και ότι εμείς θα εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα που θα υπάρξει. Τα πρώτα χρόνια το Συμβούλιο μας έλεγε ναι, καλά δεν μας αρέσει τόσο πολύ, αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε. Τη δεύτερη φορά όμως νομίζω δεν θα έχουμε το ίδιο μήνυμα. Και το τρίτο χρόνο πια που θα συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή θα υπάρξει κίνηση. Το Συμβούλιο τα γνωρίζει αυτά και γι' αυτό έκανε προσπάθειες να αποφύγει την πρόταση αυτή κανονισμού. Να μην καταλήξει δηλαδή ενώπιόν μας. Δεν είμαι λοιπόν εγώ τόσο απεσιόδοξη ό,τι αφορά την απόδοση τη προσπάθεια αυτής. Για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, εξετάζοντας το χρονοδιάγραμμα που έχουμε μπροστά μας, ανησυχώ ότι το Συμβούλιο θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο. Οχτώ χρόνια χρειάστηκε η μεταρρύθμιση της Όλαφ. Οχτώ χρόνια. Όσοι λοιπόν εγκύπτουν τώρα στην προσπάθεια αυτή θα χρειαστούν πολύ αιμονή και επιμονή μια πενταετία για μένα δεν είναι τίποτα στην, στον χρονικό αυτό ορίζοντα. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε και να συνεργαστούμε με την Όλαφ όπως αυτή είναι τώρα και να καταβάλουμε προσπάθεια να προχωρήσουν τα πράγματα. Και γι' αυτό θα σας πω το εξή για αυτό το υπερβολικό reporting που μας επισημαίνεται ότι σας επιβάλλουμε. Εμείς κάναμε προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τα σφάλματα του παρελθόντος και έχουμε 10 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και με όλες αυτούς τους εντυπωσιακού, τα εντυπωσιακά νούμερα που βλέπουμε, έχω πει πώς είναι δυνατόν ούτε ένας γενικός διευθυντής της Κομισιόν να μην έχει παρατηθεί μέχρι τώρα. Όμως δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε πλέον αυτά. Σε ορισμένε περιπτώσεις είναι δύσκολο να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα. Αν εσείς έχετε διαπιστώσει κάτι, τότε πρέπει και να λάβετε το λόγο να βγείτε να μας το πείτε. Εγώ πιστεύω πάντως ότι το σχέδιο κανονισμού που έχουμε μπροστά μας είναι καλό, θα επιτρέψει μεγαλύτερη διαφάνεια, θα προσδώσει και μεγαλύτερο κύρος στο αξίωμα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα. Ασχολούμαι πολύ με το θέμα αυτό και νομίζω ότι όντως κινείται σωστά. Και οι τροπολογίες που έχουμε καταθέσει είναι αντικείμενο κοινής διαπραγμάτευσης μαζί σας δεν σημαίνει ότι εδώ ήρθαν κάποιοι βουλευτές οι οποίοι με επιμονή προσπάθησαν να περάσουν το δικό τους. Έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά με την Όλαφ μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Έχω ωστόσο ερωτήσεις. Πρώτα, για τον Γενικό Διευθυντή που μας είπε αυτή την, για αυτή την υπόθεση Βουλγαρία-Γερμανία θα ήθελα να μάθω ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ποιοι καταδικάστηκαν στη Βουλγαρία και ποιοι καταδικάστηκαν στη Γερμανία. Ή πόσοι τέλο πάντων. Δεν γνωρίζω πολύ τίποτα για την υπόθεση αυτή και γι' αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα για τα νούμερα που είπατε. Μιλήσατε για την αύξηση της εργασία σας με το περισσότερο reporting. Ναι, αλλά εγώ διαβάζω ότι στο πιφ του Ιουλίου, στι 33 4 μου φαίνεται, ότι υπήρξε μείωση κατά 35% απέναντι στο 2011. Άρα δηλαδή κάπου υπάρχει μια εξισορρόπηση. Δεν ξέρω γιατί το, τι έγινε το 2011 και γιατί τώρα μειώθηκαν τόσο πολύ οι περιπτώσεις αυτές των αναφορών. Τώρα και μια ερώτηση προς την κυρία Μίτερμαϊερ. Έχετε δίκιο. Αυτή η υπόθεση με τους δικαιούχους δεν μας έχει ωφελήσει τα τελευταία χρόνια. Βέβαια εσείς ήρθατε εδώ στις Βρυξέλλες και κάποια εποχή, όπου, το 2007 δηλαδή, έγινε η πρώτη δημοσίευση αυτών των μεγάλων αριθμών δικαιούχων. Είναι σημαντική αυτή η ενιαία ιστοσελίδα που ζητήσατε, αλλά την έχουμε ζητήσει και εμείς. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα και σε τροπολογίες της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Και είναι και θέμα βέβαια νομικής δεσμευτικότητας της ιστορίας αυτής. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι συγκρισιμότητα με τα στοιχεία, με τα δεδομένα και της δικής σας οργάνωσης για παράδειγμα. Έχουμε ολόκληρα εντός εισαγωγικών νεκροταφεία δεδομένων κρυμμένα σε, διάφορα, σε διάφορες ε, μεριές και αυτά δεν χρησιμοποιούνται, δεν τα εκμεταλλεύεται κανείς. Τώρα, η ερώτηση του κύριου Γκάιερ και την επαναλαμβάνω και εγώ προς τον κύριο Γενικό Διευθυντή. Συνεργασία με τις χώρες μέλη. Πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε ώστε να προχωρήσει αυτή η συνεργασία και οι χώρες μέλη να βελτιώσουν σημαντικά τα, τη βάση που προσφέρουν στις εργασίες της ε, Όλαφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρέστρο. Τον κύριο Κονέριστε Γιόγκ, καλό να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο αποσκεκλημένους μας. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω αυτό το θέμα και τύπος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έχουμε μια πρώτη οδηγία της Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καταλήξουμε σε μια εναρμόνιση του ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Επίσης, θα υποβληθεί και πρόταση για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκή Αγγελική Αρχή. Ε, έχω την αίσθηση όμως ότι υπάρχουν επικαλύψεις εδώ και μία σύγχυση της κατάστασης. Ο Ευρωπαίος Αγγελέας είναι κάτι πολιτικό, ενώ η οδηγία είναι κάτι νομικοτεχνικό. Όλα αυτά μπερδεύουν κάπως τα πράγματα. Εμείς, η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, θα πρέπει να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο θέματα. Ας ξεκινήσουμε από την οδηγία. Στο Συμβούλιο έγινε εκτενή συζήτηση για τη νομική βάση το 325.4 δηλαδή τη συνθήκες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μας είπαν το 83.2 αφορά το ποινικό δίκαιο. Και μάλιστα θεωρήσαμε ότι κατάλληλη νομική βάση ήταν μάλλον το 83.2. Τελικά επιλέχθηκε άλλο άρθρο. Για το 53.4 είπα, μας είπαν ότι αφορούσε ειδικό, νο, ειδικό νόμο, lex specialis. Εγώ θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την αντίθετη επιχειρηματολογία. Ότι δηλαδή οι τρόποι εφαρμογής θα πρέπει να εμπίπτουν στο άρθρο 83 και όχι το αντίθετο. Και δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη της Όλαφ. Δεύτερον, ας υποθέσουμε ότι ένα κράτος μέλος εφαρμόζει αυτό το κείμενο έχουμε κάποια διάπραξη απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης για κονδύλια που ε, αφορούν προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα. Τι θα εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής αυτής της διατύπωσης. Μόνο τα κοινοτικά κονδύλια ή και τα μικτά κονδύλια που είναι εθνικά και κοινοτικά. Εμείς θεωρούμε ότι τέτοιου ε, προτάσεις αφορούν και τα δύο είδη ε, κονδυλίων. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίζεται αμυγός στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σε περίπτωση εφαρμογή έχουμε και εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, μια και πολλές φορές υπάρχει συγχρηματοδότηση για ένα πρόγραμμα. Τι σημασία έχει από πού πηγάζουν τα κονδύλια, αν είναι κοινοτικά ή εθνικά, όταν πρόκειται για μεικτό πρόγραμμα. Πιστεύω ότι η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι συνολική. Και θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουν μια σφαιρική προσέγγιση. Δηλαδή από κοινού τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρουν ένα επίπεδο συνεννόησης. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ελάχιστες ποινές και το θέμα της παραγραφής. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ε, προθεσμίες παραγραφής και το αξιόπινο επίσης ε, να έχει διαφορετική βαρύτητα και άρα να ισχύουν και διαφορετικές ε, περίοδοι παραγραφής. Και συμφωνώ ότι χρειάζεται κάποια αναρμόνιση των περίοδων παραγραφής. Αλλά όταν μιλούμε για ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, η πρόταση αυτή είναι ουσιαστικά ρηξικέλευτη. Πρώτη φορά έχουμε τέτοιο είδους αλλαγή σε διατάξεις ποινικού δικαίου. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να προηγηθεί η συζήτηση με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν να καταλήξουμε σε αυτή την πρόταση για τις ελάχιστες ποινές. Δεν λέω ότι είμαστε καταρχήν κατά, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να προηγηθεί η συζήτηση. Και δεν αρκεί η μία των ελάχιστων αυτών ποινών μόνο σε ένα τέτοιο ειδικό κείμενο. Σε ό,τι αφορά την εκπρόσωπο της Διεθνούς Διαφάνειας. Άκουσα με προσοχή την παρουσίασή σας και δεν καταλαβαίνω τι θέση έχει αυτό το όργανο, το εργαλείο που προτείνεται, αυτός ο μηχανισμός, στο διεθνές δίκαιο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσετε την ε, συμπερίληψη αυτού του μηχανισμού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όχι μόνο του κοινοτικού δικαίου, αλλά διεθνού δικαίου. Γιατί και οι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Μία ακόμη παρατήρηση για την ΟΛΑΦ. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ε, αρκετά ζωήρη συζήτηση και δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση την ΟΛΑΦ τότε, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει η Όλαφ να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα κοινοτικά κονδύλια του προγράμματος Ηρακλής. Γιατί αν δεν βρούμε πιο αποτελεσματική λύση για τις ερευνητικές μεθόδους της Όλαφ και αν δεν καταλήξουμε σε αποτέλεσμα για το θέμα αυτό, πώς Πιστεύω ότι θα εγκρίνουμε, μπορούμε να εγκρίνουμε αύξηση κονδυλίων ενώ δεν έχουμε προηγουμένω συνεννοηθεί για τα επιμέρου στοιχεία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων τη ΟΛΑΦ στις διάφορες έρευνες. Τώρα για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Αγγελική Αρχή. ΕΠΟ. Είναι πολύ εύκολο και απλό να λέει κανεί ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Γιατί υπάρχουν ε, πολλέ εναλλακτικέ λύσει, πολλά μοντέλα. Ο Ευρωπαίο εισαγγελέα σίγουρα θα πρέπει να συνεργαστεί με τι εθνικέ εισαγγελίε, εθνικέ εισαγγελικέ αρχέ. Τώρα, αν θα αποτελεί όντω προστιθέμενη αξία, αυτό είναι συζητήσιμο. Αν έχουμε ένα είδο ευρωπαϊκού FBI με άμεσε ανακριτικέ αρμοδιότητε, ναι, θα υπάρχει προστιθέμενη αξία. Όχι όμω όταν απλώ προλέβουν υποχρεωτική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εθνικών εισαγγελιών. Είναι πολύ εύκολο να λέτε ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση, η ιδανική λύση και θα λυθούν όλα τα προβλήματα σαν είναι πανάκια. Θα εξαρτηθεί τι ειδικά χαρακτηριστικά θα έχει αυτή η πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Και παραλαμβάνω ότι η Εθνική Εισαγγελή είναι κατά τη ε, ε, ίδρυση μια τέτοια μιας τέτοιας ε, πανευρωπαϊκής αρχής. Οπότε έχω κι εγώ πολλά ερωτηματικά. Γιατί οι εθνικοί Εισαγγελεί δεν ενδιαφέρονται η Όλαφ ενδιαφέρεται, η διεθνής ε, διαφάνεια ενδιαφέρεται. Γιατί όμω η Εθνική Εισαγγελία είναι κατά τη πρόταση. Ευχαριστώ. Σα ε. Σας ευχαριστώ κύριε Διόγκ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σκυλακάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα ζητώ συγγνώμη γιατί είμαι σκιώδης συγητής και ήμουν στην ΕΚΟΝ, έτσι δεν μπόρεσα λοιπόν να είμαι από την αρχή της πολύ σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας. Πρώτα θα ήθελα να πω ότι η απάτη και η διαφθορά είναι πολύ πιο ευρύτερα, πολύ ευρύτερα διαδεδομένες από ό,τι καν τολμούμε να το διανοηθούμε. Πρόκειται για κάτι που έχει τρομερή διάδοση και σε άλλους τομείς αλλά και στην οικονομική πολιτική. Δεν μπορούμε να μιλούμε για δημοσιονομική ένωση όταν το χρήμα τελικά τυχαίνει πολύ διαφορετική μεταχείρισης στα διάφορα μέρη της Ένωσης. Χρειαζόμαστε και μία ένωση κατά της διαφθοράς. Δεν θα μπω βέβαια σε λεπτομέρειες τώρα, θα πω μόνο ότι γνωρίζουμε από την διεθνή διαφάνεια, από την έκθεση της διεθνούς διαφάνειας για τις δωροδοκίες δημοσίων αξιωματούχων των χωρών μελών όπου μάλιστα υπάρχει και ένας αριθμός δημοσκοπήσεων σε όλο τον κόσμο αλλά και στις χώρες μέλη. Έχουν ρωτήσει δηλαδή τον κόσμο αν δωροδόκησαν κάποιους ή αν οι ίδιοι δωροδοκήθηκαν. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και τομείς και χώρες και περιφέρειες όπου είναι ευρύτατα διαδεδομένο το λάδωμα. Και προφανώς εφόσον υπάρχει δωροδοκία για παράδειγμα κάποιων τελωνιακών αρχών στην Ένωση ασφαλώς φύγονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Δεν φαντάζομαι να αναμένει κανείς ότι όταν κάποιος δωροδοκείται, κάποιος δηλαδή που χειρίζεται χρήματα των φορολογμένων, θα έχει περισσότερες τύψεις συνειδήσεως εφόσον καταχραστεί χρήματα των Ευρωπαίων φορολογμένων. Αντίθετα μάλιστα θα το κάνει περισσότερο αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από την ε, διεθνή διαφάνεια περισσότερα για τις δημοσκοπήσεις αυτές όπου πραγματικά μπορεί κανείς να θέσει τον δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων διότι δεν μιλούμε εδώ για διαφθορά που θεωρούμε ότι υπάρχει είναι πραγματική διαφθορά και οι άνθρωποι μιλούν ελεύθερα διότι πρόκειται για μικρού, μικρής κλίμακας διαφθοράς και πολύ συχνά βέβαια οι άνθρωποι μιλούν ελεύθερα γιατί δεν γνωρίζουν ποιο είναι αυτός που του παίρνει τη συνέντευξη δεν τον βλέπουν προσωπικά δηλαδή. Και θέλω να μάθω επίσης αν έχουν διασυνδέσει καμιά φορά αυτού του είδους τις δωροδοκίες με την απάτη σε βάρος του ευρωπαϊκού χρήματος ή αν έχουν χρησιμοποιήσει πάλι διεθνείς διαφάνεια δηλαδή ε, τις ε, τεχνικές αυτές για να μετρήσει την διαφορά. Διότι γνωρίζουμε ότι συλλαμβάνουμε και μάλιστα μόνο κατά τύχη θα έλεγα, εγώ ψαρεύουμε κάποια μικρά ψαριά της διαφθοράς. Είναι τα δίχτυα μας τόσο αναποτελεσματικά που μόνο κατά τύχη μεγάλη μπορεί να πιάσουμε κάτι. Τώρα θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κέσλερ για ένα που, θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Πόσες έρευνες της Όλαφ γίνονται από δική της πρωτοβουλία και πόσες διεξάγονται μετά από κάποια καταγγελία. Διότι εάν, όπως υποψιάζομαι, άλλωστε το έχουμε ξανασυζητήσει παλαιότερα, αν ισχύει το ότι περίπου 90% των ερευνών μας γίνονται διότι κάποιος έχει καρφώσει ή έχει καταγγείλει, αυτό σημαίνει ότι εφόσον υπάρχουν διεφθαρμένα συστήματα τα οποία κρατούν κλειστό το στόμα των ενδιαφερομένων, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να παρέμβει το ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν δηλαδή δεν έχουμε έρευνε ίδιας πρωτοβουλία και μάλιστα θα έλεγα που να καλύπτουν το 50% των υποθέσεων που χειρίζεται η Όλαφ, όπου να μπορούν οι δυνάμεις της Όλαφ να παρέμβουν σε τομείς όπου γνωρίζουμε ότι υπάρχει διαφθορά αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, τότε δεν πρόκειται να εμπνεύσουν κανένα φόβο ε, στους ανθρώπους οι οποίοι κλέβουν τα ευρωπαϊκά χρήματα. Και αυτό πολιτικά είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή νότια, βόρεια, ανατολικά, όλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Είτε διότι καλούνται να ενισχύσουν άλλες χώρες, είτε διότι αντιμετωπίζουν βαριά προγράμματα λιτότητας. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν γίνει πια πολύ ευαίσθητοι στο θέμα αυτό. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μας ενώνει ενώνει τους ευρωπαϊκούς λαούς ο αγώνας κατά της διαφθοράς, περισσότερο από ποτέ. Και νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε πολύ περισσότερο θάρρος και πολύ περισσότερη πρωτοβουλία. Και ας μην φοβούμαστε να μιλήσουμε για το ε, γραφείο του Ευρωπαίου Αγγελέα, την Όλαφ και όλα τα άλλα συναρμόδια όργανα να, να έχουν αυτό να γίνει ένα ευρωπαϊκό FBI. Το αμερικανικό FBI έχει υπάρξει ιδιαίτερα επιτυχές για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου κλίματος και στα τελευταία 100 χρόνια μάλιστα, 90 τέλος πάντων, 90 χρόνια πέστε. Πρέπει λοιπόν τουλάχιστον να το συζητήσουμε, διότι στην πραγματικότητα έχουμε αποτύχει. Και μάλιστα εγώ θα ήθελα να διεξαχθεί συζήτηση, και τελειώνω εδώ, ελπίζω να μην μακρηγόρησα πολύ, για τις εκθέσεις του ΟΣΑ, για τις δωροδοκίες ξένων αξιωματούχων. Αν διαβάσετε τις εκθέσεις αυτές θα δείτε ότι ακόμη και σε ε, δικαιο... Ε, δικαιικά συστήματα που λειτουργούν καλά υπάρχει σημαντικότατη διαφθορά, δωροδοκίες δηλαδή αξιωματούχων σε άλλες τρίτες χώρες. Και οι περισσότεροι τελικώς, τελικώς διαφεύγουν τη δίωξη, ενώ αυτοί που έχουν κάνει τις, ε, έχουν κάνει τις δωροδοκίες. Το πολύ πολύ με ένα ελαφρό χτύπημα στον νόμο. Ενώ βλάπτονται βαρύτατα τα συμφέροντα των χωρών όπου ε, είναι ο δωροδοκούμενος αξιωματούχος. Και αν δεν, δεν υπάρχει, αν δεν υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από τις χώρες οι οποίες τέλος πάντων έχουν καταφέρει καλύτερα να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, τι να περιμένουμε τότε από τους υπολείπους, από τις υπόλοιπες χώρες, όπου οι άνθρωποι είναι πιασμένοι στην παγίδα της συστημικής διαφοράς, διαφθοράς συγγνώμη, και του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστώ κύριε Σκυλακάκη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πολ Ρούμπιχ και μετά στην κυρία Μέλη Αντερστότερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμένα εν προκειμένου με ενδιαφέρει τι μπορεί να γίνει προληπτικά. Έχουμε και τη διαδικασία reverse charge για τον φόρο προσθέμενης αξίας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να μειωθούν οι απάτες ε, στον τομέα του φόρου προσθέμενης αξίας. Από την άλλη μεριά έχουμε για παράδειγμα στα Ηνωμένα Εμμυράτα ζώνες ελεύθερες φορολογίας, όπου εκεί διεξάγονται πολλές συναλλαγές. Αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις στον έλεγχο των απατών. Ευχαριστώ κύριε Ρουμπίκ. Η κυρία Άντερς Ντότερ. Um, Εγώ πρώτα ευχαριστώ την κυρία Μάιερ για την παρουσίασή της. Εμείς υποστηρίζουμε πολύ την έκθεση της για τους whistleblowers, αυτούς δηλαδή που καταγγέλουν στις αρχές πράγματα που κάνουν συνάδελφοί τους. Τώρα έχουμε και τα θέματα ε, από την Συμφωνία Καπνού. Γνωρίζουμε και με τις, ε, από τις συζητήσεις στη Γενέβη ότι το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού γίνεται όλο και μεγαλύτερο και ανακατεύεται πλέον και σε πολιτικές συζητήσεις. Στο γραφείο μου εμείς εξετάσαμε τις συμφωνίες για τον καπνό και διαπιστώσαμε πολλά μέτρα σχετικά με το τι είναι παραποιημένα τσιγάρα όπου εκεί συλλέγονται εισφορές στα σύνορα και εκεί γίνονται περισσότερο εκστρατείε για την καταπολέμηση των παραποιημένων τσιγάρων και όχι του λαθρεμπορίου τσιγάρων, πραγματικών τσιγάρων δηλαδή. Εγώ βρίσκω ότι το θέμα είναι περισσότερο πολιτικό και λιγότερο επιχειρησιακό για την Όλαφ τώρα, αλλά ποια αποτελέσματα αναμένει η Όλαφ από το ανακάτεμα όλων αυτών τώρα, δηλαδή της ε, παρεμπόδισης του λαθρεμπορίου παραποιημένων τσιγάρων σε σχέση με την ε, πάταξη του λαθεμπορίου ε, αληθινών σιγάρων και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Μια ναι, και δεν ε, ζητάει άλλος κανείς το λόγο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Τζοβάνι Κέσλερ για να απαντήσει πρώτες ερωτήσεις και μετά στην κυρία Γιάννα Βέτερμάγερ. Καταρχήν, η ερώτηση που τέθηκε στον κύριο Κέσλερ από τον εισηγητή μας τον κύριο Γιάννη Γκάιερ είναι η εξής. Κατά τη γνώμη σας, Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες αυτής της ε, Ευρωπαϊκής ε, εισαγγελία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις που υποβάλλατε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τις ε, πολλές και διάφορες ερωτήσεις που τέθηκαν για το ΕΠΟ, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή στα, είχα καταρχήν 10 λεπτά χρονομιλίας, ε, μίλησα 20 λεπτά και δεν μπόρεσα να τα καλύψω ούτε μέσα 20 λεπτά όλα. Γι' αυτό σας ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, γιατί μέσα στα 3 λεπτά που έχω τώρα είναι αδύνατο να καλύψω όλες τις λεπτομέρειες για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία άλλη φορά να επανέλθουμε πιο διεξοδικά στο θέμα. Ζητώ συγγνώμη γιατί θα απογοητεύσω πολλούς με αυτή την πραγματικά επιγραμματική μου απάντηση. Για τις ε, αρμοδιότητες. Βρισκόμαστε, όπως είπα, σε προκταρκτική φάση. Δεν έχουν ε, προσδιοριστεί όλες οι αρμοδιότητες. Πάντως, ε, με βάση αυτό που προβλέπει και η συνθήκη, μιλούμε για εγκλήματα που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, α, ε, μιλούμε ουσιαστικά για τις τωρινές αρμοδιότητες της ΟΛΑΦ ή για εγκλήματα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογή που αναφέραμε για τη σύγκληση ή την εναρμόνιση των ε, ποινικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση την πρόταση δηλαδή που μόλις τον περασμένο Ιούλιο υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ξέρετε, οι συνθήκες προβλέπουν ότι σε ένα μεταγενέστερο στάδιο και αν συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Αυτή είναι δυνατότητα όμως μπορεί να ξεπηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Αρχικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει αρμοδιότητα για εγκλήματα που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή απάτη, διαφθορά, λαθρεμπόριο, γιατί είναι θέματα που επηρεάζουν ε, και τα έξοδα της δαπάνης αλλά και την απώλεια εσόδων. Τίποτα καινούργιο λοιπόν αυτή την άποψη. Αλλά παρόλα αυτά θα σημαίνει ένα βήμα προόδου η ίδρυση του ΕΠΟ. Ε, για το ίδιο θέμα, συμφωνώ με μερικούς από εσάς, μπορώ να αναφερθώ τώρα ονομαστικά στον καθένα, ζητώ συγγνώμη, αλλά προσπάθησα να συγκεντρώσω τις ερωτήσεις ανά θέμα. Ποιο μοντέλο θα προτείνουμε. Φυσικά, το μοντέλο θα είναι σημαντικό, αλλά το ΕΠΟ, η Ευρωπαϊκή Συγγελία, δεν είναι μόνο ένα όνομα. Και και στις συναντήσεις μας με τις εθνικές αρμόδιες αρχές αλλά και με τους ε, όλους τους ε, Γενικούς Εισαγγελείς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε και τον περασμένο ήταν την πρόσφατη με τους εισαγγελείς ήδη είχαμε πολλές ε, συσκέψεις και με τους ε, Γενικούς Εισαγγελείς και έχουμε τακτικές επαφές και μπορώ να σας διαβεβαιώσω κύριε Ντεγιόγκ ότι είμαι πολύ πιο αισιόδοξο από εσά για την αποδοχή που θα έχει πρόταση αυτή από τις εθνικές εισαγγελίες. Έχουμε λοιπόν ένα μοντέλο αυτή τη στιγμή που είναι ουσιαστικά ένα συνδυασμό ε, του κεντρικού εισαγγελικού γραφείου και των ε, εθνικών διοκτικών αρχών για την πάταξη της απάτης. Έχουμε ουσιαστικά ένα δίκτυο στο οποίο θα συνεργάζονται οι εθνικές και η Ευρωπαϊκή Αρχή. Αυτές ε, αυτοί οι εισαγγελείς θα εμπίπτουν στις εθνικές ε, εισαγγελίε, αλλά όταν χειρίζονται τέτοιου είδους εγκλήματα θα ασκούν τις αρμοδιότητες τους υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία. Σε ένα ευρύτερο δηλαδή πανευρωπαϊκό πλαίσιο υπό την ευθύνη, ε, την αιγίδα για το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής. Και αυτό που θα κάνουν η Εθνική Εισαγγελή έχει μια πανευρωπαϊκή εμβέλεια η δράση τους σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε θα έχουν και πιο ενισχυμένες αρμοδιότητες και πιο αποτελεσματική ε, έρευνα, γιατί θα ξεπεράσουμε την ε, κατάσταση του κατακαιρματισμού που έχουμε σήμερα και που μας οδηγεί σε αναποτελεσματικές έρευνες. Αυτά ως προς το ΕΠΟ, αλλά ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία για πιο λεπτομεριακή και εκτενή ανταλλαγή απόψεων, όποτε το κρίνεται σκόπιμο, ακόμη και πριν την επίσημη υποβολή της πρότασης που θα γίνει τον Ιούνιο. Είμαι στη διάθεσή σας ανα πάσα στιγμή και εγώ και η κυρία Λεμπάιχ, η αρμόδια Γενική Διευθύντρια της ε, Διεύθυνσης ε, Δικαιοσύνης, για συμμετοχή σε συζήτηση για το θέμα αυτό. Τώρα, για, το, για την αναθεώρηση του 1073. Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη αναθεώρηση. Πιστεύω ότι έχει οριμάσει η συζήτηση και βρισκόμαστε στα πρόθυρα της έγκρισης ε, της μεταρρύθμισης ε, του κανονισμού 1073 και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό γιατί θα εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια, πολλά θετικά στοιχεία και ουσιαστικά ήδη από την πρώτη Δευτέρου, από την πρώτη Δευτέρου ε, ευθυγραμμιζόμαστε με τις αλλαγές και γι' αυτό ελάχιστα θα αλλάξουν στις ε, διαδικασίες της ΟΛΑΒ, γιατί ήδη έχουμε προσαρμοστεί στις νέες διαδικασίες ε, γνωρίζοντας ποια θα είναι η μορφή του τελικού κειμένου. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα έχουν ε, τα 30% περισσότερων ε, καταγγελιών. Η περικοπή των, ε, του προσωπικού, των ανθρώπινων πόρων, όχι των οικονομικών πόρων. Ακόμη και αν έχω περισσότερα κονδύλια, τι να τα κάνω αν δεν μπορώ να προσλάβω υπαλλήλου ή αν βρεθώ με λιγότερους υπαλλήλου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα έχουμε λιγότερο προσωπικό. Επίσης, περισσότερες υποχρεώσεις, περισσότερες υποχρεώσεις και όχι επιπλέον ερευνητικέ αρμοδιότητες. Ο τίτλος της ε, δημόσια αυτής ακρόαση είναι «Οι επιπτώσεις στο ερευνητικό έργο τη ΟΛΑΦ και το συνδυασμένο αποτέλεσμα όλων αυτών των παραγόντων, γιατί ε, δεν είστε εσείς υπεύθυνοι για όλους αυτούς τους παράγοντες, αλλά εγώ τους προβλέπω ήδη και αν τους συνδυάσω, πιστεύω ότι είναι εύκολο να καταλήξουμε και εσείς και εγώ στο συμπέρασμα ότι θα έχουν πραγματικά τεράστιο αντικτύπο και μάλιστα αρνητικό ο συνδυασμό όλων αυτών των ε, παραγόντων. Ε, λιγότερο προσωπικό, ε, περισσότερο διοικητικό έργο, περισσότερη υποχρέωση ενημέρωση υποβολής εκθέσεων και περισσότερες καταγγελίες, θα έχουμε μάλλον αρνητικό αντικτύπο στο ερευνητικό έργο της Όλαφ. Ελπίζω να μην είναι καταστροφική η κατάσταση. Δεν θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε τελικά, αλλά αν με ρωτάτε ποια θα είναι η επίπτωση των μεταρρυθμίσεων στο ερευνητικό έργο, πιστεύω ότι θα είναι αρνητική. Τώρα, κάποιος ρώτησε πώς ε, έχετε περισσότερες πληροφορίες αφού οι κοινοποιήσει ε, με βάση τη σύμβαση PIF για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των κοινοτήτων μειώνονται. Κάθε χρόνο οι κοινοποιήσει που γίνονται από τα κράτη-μέλη μέσω της σύμβασης αυτής ε, αφορούν υπόνοιες ατασταλιών ή απατών. η Όλαφ είναι διαχειριστή ουσιαστικά, συγκεντρώνει όλα αυτά τα δεδομένα από τα κράτη-μέλη και προσπαθούμε να ενοποιήσουμε τα κριτήρια. Αυτό κάνει μόνο η Όλαφ. Και δεν έχει κανένα σχέση με το ερευνητικό έργο της Όλαφ. Εδώ μιλούμε για κοινοποίηση των υπονοιών ε, των κρατών μελών για απάτες και διαφορές. Όταν είπα ότι θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες καταγγελίες για διαφθορά και απάτη, όταν είπα θα αυξηθούν αυτές κατά 30%, εννοούσα τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από ε, κοινοτικά θεσμικά όργανα, από τα κράτη-μέλη, από ε, αρμόδιες αρχές, κυβερνητικούς φορείς, ε, δικαστικούς, αστυνομικούς, εξωτερικούς ελεγκτές. εκείνοι κάνουν κάποιες καταγγελίες και μας ζητούν να ξεκινήσουμε έρευνα Επίσης αναφερόμουν και σε πληροφορίες από ιδιώτες, γιατί ο κάθε πολίτης, η κάθε επιχείρηση, ο κάθε φορέας εντός εκτός Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, δίνεται να αποταθεί στην ΟΛΑΦ και να ε, καταγγείλει πιθανές ατασταλίες ή παραβάσεις, παπάτες κτλ. Κάθε χρόνο έχουμε όλο και περισσότερες τέτοιες καταγγελίες. Φέτος είχαμε 30% περισσότερες. Είναι πολλέ για να τι χειριστούμε. Αλλά καλό αυτό. Δείχνει ότι όλα γίνεται πιο γνωστή και φυσικά φαντάζομαι ότι έχουμε και εμείς περισσότερη εμπιστοσύνη, περισσότερη αυτοπεποίθηση. Τώρα αναλύουμε εις βάθος όλες αυτές τις καταγγελίες και έχουμε τις πληροφορίες στην ετήσια μας έκθεση. Από τα θεσμικά, τα κοινωτικά θεσμικά όργανα έχουμε λιγότερες πληροφορίες. Από τον ιδιωτικό τομέα έχουμε όλο και περισσότερες καταγγελίες. Οπότε αυτή η αύξηση μεγάλη οφείλεται περισσότερο στις καταγγελίες που λαμβάνουμε από ιδιωτικές πηγές παρά από τους δημόσιους φορείς. Και αυτό κάτι δείχνει βέβαια, θα, θα αναλύσουμε την κατάσταση και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Πάντως δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του το, τι κοινοποιούν τα κράτη-μέλη μέσω της σύμβασης ε, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και των πληροφοριών ή των καταγγελιών που λαμβάνει η ΟΛΑΦ. Πολλές φορές ο κόσμος μπορεί να μην έχει ε, εμπιστοσύνη στις εθνικές αρχές και να προτιμά να κάνει τις καταγγελίες απευθείας στην ΟΛΑΦ. Μερικές φορές οι εθνικές αρχές ε, κάνουν καταγγελίες λέγοντας ότι αυτό το, το έγκλημα μας ξεπερνά, ξεπερνά τις αρμοδιότητές μας, είναι πολύ περίπλοκο, βοηθήστε μας και αυτό εύλογο είναι. Και πολύ συχνά και εμείς εθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να μα υποβάλουν πιο συχνά καταγγελίες πληροφορίε. Δεν είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερε πληροφορίε, αντίθετο, γιατί κατακλυζόμαστε από πληροφορίε, αλλά θέλω, θέλουμε να ενισχύσουμε τι συνεργασίε μεταξύ των αρμοδίων αρχών και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Και έρχομαι εδώ και στο θέμα του κυρίου Σκυλακάκη. <laughs> Είναι ο, ο μόνος τον οποίο αναφέρομαι ονομαστικά, <laughs> συγγνώμη γιατί είσαι τελευταίο και θυμάμαι καλύτερα. Τώρα, με ρωτήσατε τι κάνει η Όλαφ από τις έρευνες. Ένα μικρό τμήμα των δικών μας ερευνών γίνονται με δική μας πρωτοβουλία. Πάντως στον κανονισμό 1073 διαβάζω και φαντάζομαι θα το εφαρμόσουμε αυτό ότι πρέπει να ξεκινήσουμε έρευνες όταν έχουμε επαρκώς σοβαρές υπόνοιες Δηλαδή, τα τρία S, sufficiently serious suspicions, επαρκώς σοβαρ, ε, επαρκείς και σοβαρές υπόνοιες. Αν περιμένουμε να έχουμε επαρκείς και σοβαρές υπόνοιες, μπορούμε να περιμένουμε και να μην ξεκινήσουμε ποτέ μια έρευνα. Με την αναθεώρηση του 1073, ένα από τα τρία S τα διαγράφηκε, καλό αυτό, αρκούν επαρκείς υπόνοιες αυτό το θεωρούμε αρκετά σοβαρό, ώστε να διαγράψουμε το σοβαρό. Δηλαδή έμειναν σας πίσω. Το Σύριος διαγράφηκε. Αλλά ήδη έχουμε 1.300 πληροφορίες καταγγελίες το χρόνο. Εγώ δεν είμαι σε θέση με την έλλειψη προσωπικού και με, όλα, με όλους τους λόγους που σας ανέφερα να βγω και να ψάχνω για περισσότερες πληροφορίες. Και επιπλέον από την 1η Φεβρουαρίου θα δούμε, μπορούμε να δίνουμε μέσα σε δύο μήνες απάντηση για το αν θα ξεκινάει ή όχι μια έρευνα. Προηγουμένως, πριν την αναθεώρηση του κανονισμού, η προθεσμή για την απόφαση αυτή ήταν ε, κατά μέσο όρο 7 μήνες. Τώρα κατά μέσο όρο θα είναι 1,1 μήνας. Οπότε αυξήθηκε η ταχύτητα ο 1073 μας λέει τώρα ότι μέσα σε δύο μήνες πρέπει να λαμβάνουμε την απόφαση για το θα ξεκινάει όχι μια έρευνα. Έχουν αλλάξει πολλά στις εσωτερικές διαδικασίες, έχει γίνει μια απλούστευση και πραγματικά το προσωπικό δουλεύει άοκνα και σκληρά και τα καταφέρουμε. Και επίσης έχουμε και κόσμο που μπορεί να ε, αναστεί πληροφορίες. Εγώ ούτε στα πιο φιλόδοξα μόνιρα δεν ε, ονειρευόμουν να γίνω Έντγκαρ Χούβερ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό κάτι τέτοιο. Ίσως γιατί δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι θέμα μόνο χαρακτήρα. Δεν έχω ούτε προσωπικό, ούτε υπαλλήλου και δεν έχω και καν τη νομική βάση, ούτε και τι εξουσίε και τι αρμοδιότητε για κάτι τέτοιο. Αν μου το ζητήσετε, πολύ ευχαρίστω. Ξέρω πώ ε, λειτουργεί ε, το FBI. Έχω κάποια εμπειρία και έχουν και κάποιε επιχειρήσει undercover. Εμεί πώ θα το κάνουμε. Εγώ δεν μπορώ καν να πάω να ανοίξω, ένα, να, ε, να ανοίξω έναν τραπεζικό λογαριασμό. Τι έρευνα να κάνουμε αν δεν έχουμε μια τέτοια πρόσβαση που είναι το, το α, το πιο απλό πράγμα η πρόσβαση σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάμε κάποιες έρευνες και με δική μας πρωτοβουλία, θα ήταν η ερώτηση, όταν έχουμε υπόνοιες, όταν έχουμε υποψίες ότι σε εθνικό επίπεδο δεν επιλαμβάνεται η αρμόδια αρχή. Και το διαβάζουμε και σε εφημερίδες. Μερικέ φορέ μα στέλνετε τι πληροφορίε. Μερικέ φορέ τι διαβάζουμε εμεί. Έχουμε τι ε, κοινοβουλευτικέ ε, ερωτήσει που επισημαίνουν επίση κάποια θέματα. Λέμε, α, ενδιαφέρον και αυτό. Μετά κάνουμε τον έλεγχο σε εθνικό επίπεδο, βλέπουμε ότι τίποτα δεν γίνεται, οπότε τότε με δική μας πρωτοβουλία ξεκινάμε. Λίγες όμω έρευνε έτσι. Και άλλη δυνατότητα δεν έχουμε με την παρούσα νομική βάση και με τους ανθρώπινους πόρους που έχουμε. Ούτε με την αναθεώρηση θα αλλάξει ριζικά η κατάσταση. Η έρευνε με δική μας πρωτοβουλία είναι πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των ερευνών μας. Πάντως πιστεύω ότι αν η Όλαφ λειτουργεί σωστά και αυτό επιδιώκουμε, αν καταφέρει να δώσει μια απάντηση σε ένα έφθετο χρονικό διάστημα, έστω και με λιγότερο προσωπικό, πιστεύω ότι και ο κόσμος και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, αν δώσουμε την εντύπωση ότι όχι εμείς είμαστε οι ταραχοποιοί, όχι Παναγίτσα μου ήρθε η Όλαφ και μου χτυπάει την πόρτα, αλλά ότι είμαστε ένα σημαντικό σφορές των κοινοτικών θεσμικών οργάνων για να λύσουμε ένα πρόβλημα, και είμαστε ένα του, τότε πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες, όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά καλύτερες. Και έτσι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε καλύτερα και στην αποστόλη μας. Θεωρώ ότι μία αποτελεσματική πάταξη της απάτης και της διαφθοράς εντός των κρατών μελών και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων ε, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να γίνεται από κοινού δεν είναι να πάει και να χώνει τη μύτη μη της παντού η Ολάφ με τους κατασκόπους της που δεν έχει τόσοι άλλος. Το θέμα είναι, είναι μια ομαδική εργασία. Θα πρέπει να γίνεται με συνεργάσιμο πνεύμα και θα πρέπει οι να, γίνονται, να δίνονται με εντυμότητα, με εμπιστοσύνη και με ειλικρίνεια. Αν επιμερίσουμε αυτό το έργο και ο καθένας ανάλογα με τις ευθύνες του αναλάβει το δικό του τμήμα, εμείς κάνουμε τις έρευνες, αλλά αυτοί που δουλεύουν και βλέπουν ε, τις ατασταλίες να τις ε, ε καταγγέλουν. Αν έχουμε λοιπόν κοινέ αξίες και εμπιστοσύνη αμοιβαία, είμαι αισιόδοξο ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά είναι συλλογικό το έργο, δεν είναι ατομικό. Τώρα, δύο λόγια για την οδηγία σε ό,τι αφορά το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο. Τώρα δεν πρόκειται να συζητήσουμε το θέμα της νομικής βάσης. Αν δεν κάνω λάθος, η νομική βάση είναι το άρθρο 325. Θα γίνει διεξοδική συζήτηση ε, στις νομικές υπηρεσίες για τη νομική βάση. Αλλά έχουμε την ίδια τη συνθήκη της Λισαβόνας και αυτό που κάνουμε σήμερα δεν είναι διαφορετικό από αυτό που ισχύει με βάση τη σύμβαση. Τη σύμβαση του 95 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ε, κοινότητας, την ΠΙΦ, που δεν την έχουν υπογράψει όλοι, αλλά όπως λέμε, την λισαβονοποίησαμε, όπως λέμε στην κοινοτική ορολογία. Έχουμε πια την συνθήκη της Λισαβόνας, εντάξαμε την σύμβαση αυτή της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων, όχι της κοινότητας, αλλά της Ένωσης, δεν είναι πια τρίτος πυλώνας, έχει ενταχθεί στη συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί πρωτογενές δίκαιο και υποχρέωση για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτά ως προς την νομική βάση, αλλά σίγουρα θα γίνει σχολαστική συζήτηση και ανάλυση από τις νομικές υπηρεσίες. Πάντως είναι σημαντικό να γίνει η συζήτηση αυτή για να καταλάβουμε όλοι ποιο είναι το νέο πλαίσιο με βάση τη συνθήκη της για τη δικαιοσύνη. Γιατί προηγουμένως η δικαιοσύνη ήταν κάτι ξεχωριστό δεν είναι στην συνθήκη. Τώρα μετά τις ειδικές της και η δικαιοσύνη, το μέσο δικαιοσύνη εμπίπτει στις αρμοδιότητες της κοινότητας. Τώρα, κύριε Δε Γιόγκ, ελάχιστες ποινικέ κυρώσεις. Παρακαλώ, προσοχή. Ουδέποτε δεν είπαμε ελάχιστες ποινές, ελάχιστες καταδίκες. Ίσως εκεί ήταν η παρεξήγηση. Δεν ξέρω πώς θα το πω καλά στα αγγλικά, αλλά είπαμε ε, ελάχιστες ποινές. Τώρα, μπορεί η, μετά την εκδίκηση απόφασης ε, οι ποινές είναι ακόμη χαμηλότερες ανάλογα με ελαφρυντικά ίσως που θα ληφθούν υπόψη ηλικία κτλ. Αλλά μερικές χώρες δεν, δεν τις έχουν ακόμη. Λίγες είναι οι χώρες βέβαια που δεν έχουν καθόλου κάτι τέτοιο και θα είναι καινούριο για αυτές. Αλλά μια και μιλούμε για τα κοινοτικά κονδύλια, δεν είναι μόνο Ολλανδικά, Ιταλικά, Γερμανικά. Είναι τα κοινά κονδύλια και μια και οι εγκληματίες είναι οι ίδιοι. Αν γνωρίζουν οι εγκληματίες ότι δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν την επική νομοθεσία μιας χώρας, με το ελάχιστο που προτείνουμε για έξι μήνες για την παραγραφή, ή μάλλον όχι για την ποινή, σε μερικές περιπτώσεις θα είναι ακόμη χαμηλότερη ποινή. Δεν νομίζω ότι είναι καμιά φοβερή επανάσταση και μπορούμε εύκολα να την εφαρμόσουμε. Και τέλος, εκπρόσωπος των Πρασίνων, αν δεν κάνω λάθος, έθεσε μία ερώτηση εμείς προσπαθούμε και πιστεύω ότι τα καταφέρουμε να μην μπερδεύουμε το θέμα της παραποίησης των σιγαρέτων με το λαθρεμπόριο σιγαρέτων ή προϊόντων καπνού. Δεν πρόκειται εδώ να προστατεύσουμε συμφέροντα εμπορικά ή άλλα, αλλά τα σεβόμαστε. Εμείς πάντως είμαστε αρμόδιοι για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττονται και από το λαθρεμπόριο και από την παραποίηση των προϊόντων, από τα πλαστά προϊόντα. Εσείς αναφερθήκατε στα προϊόντα καπνού. Στην περίπτωση αυτή, στον τομέα του καπνού, είναι αλληλένδετα το λαθρεμπόριο με την παραποίηση. Τα σιγαρέτα λαθρεμπορίου μπορεί να είναι ε, σιγαρέτα που δεν είναι μάρκας, ή να είναι παραποιημένα ή να είναι αυθεντικά προϊόντα μεγάλο, μεγάλο, σημαντικού εμπορικού σήματος, χωρίς που δεν έχουν παραποιηθεί, που όμως στη συνέχεια μέσω λαθρεμπορίου κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Έχουμε τρία διαφορετικά είδη. Και εμείς τα λαμβάνουμε όλα υπόψη, τα αντιμετωπίζουμε όλα, γιατί είναι οι ίδιοι εγκληματίες αυτοί που είναι οι λαθρέμποροι που χωρίς να πληρώνουν τελωνιακούς δασμούς διακινούν επώνυμα σιγαρέτα ή παραποιημένα ή σιγαρέτα που δεν είναι μάρκας και που κυκλοφορούν λαθρέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Η ΟΛΑΦ τις αντιμετωπίζει όλες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ετέθησαν σαφείς ερωτήσεις από την κυρία Γκρέσλερ και την κυρία Γιόγκ. Η κυρία Γκρέσλε ρώτησε στην περίπτωση της διαφθοράς ποια ήταν η απόφαση του γερμανικού και του βουλγαρικού δικαστηρίου. Ο κ. Ντε ρώτησε ποιε είναι οι στάσεις έναντι διαφθοράς όπου υπάρχει μεικτή χρηματοδότηση, δηλαδή ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση. Ε, ποια προσέγγιση ακολουθείτε σε αυτή την περίπτωση. Απάντηση προς την κυρία Γκρέσλε. Διαβάζοντας την έκθεσή μας, βλέπετε ότι είναι γνωστό ότι εκείνοι που το διέπραξαν το αδίκημα αυτό στη Γερμανία καταδικάστηκαν εδώ και πολλά χρόνια. Ε, το άτομο που ερευνά του στην Βουλγαρία ε, έλαβε ποινή 12 ετή για πολλά εγκλήματα που διέπραξε το πρωτοδικείο, το πρωτοδικείο στην Βουλγαρία και πριν από μερικές μέρες από το εφετείο αθώθηκε. Και δεν τελείωσαν τα πράγματα διότι οι διοκτικές αρχές πιθανότατα θα πάνε σε ανώτατο δικαστήριο. Οπότε ε, θα σας ενημερώνω. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της περασμένης εβδομάδας. Δεν έχει σημασία αν είναι βουλγαρική υπόθεση ή γερμανική υπόθεση. Έχουμε πολλές τέτοιες υποθέσεις. Νομίζω ότι απάντησα το ερώτημα. Όσον αφορά την οδηγία όσο έχει και τις αρμοδιότητες της Όλαφ, αν έχουμε σε μια κρατική προμήθεια 1% ευρωπαϊκά χρήματα, έχουμε αρμοδιότητα να επιληφθούμε. Αν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά χρήματα, δεν έχουμε την αρμοδιότητα. Το ίδιο θα ισχύει και για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και την εφαρμογή της οδηγίας. Δεν ξέρω αν συμπεριλαμβανόταν αυτό που λέω στο ερώτημα, αλλά σε κάθε κράτος μέλος αν εγκριθεί η οδηγία όπως ε, ελπίζω για το συστικό δίκαιο. Και υπάρξει περίπτωση διαφθοράς ε, σε, ένα διαγωνισμό για προμήθεια. Και δεν υπάρχουν όμως οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Αυτό θα είναι θέμα που θα διευθετείται αποκλειστικά από την, ε, από, τον εθνικό, από την εθνική ποινική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους. Αν έχουμε 0,1% έστω χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσης που εμπλέκονται στην υπόθεση θα είναι κάτι που θα διευθετείται από το εθνικό δίκαιο εναρμονισμένο με την οδηγία. Οπότε για το ίδιο αδίκημα που έχει διαπραχθεί σε μια χώρα μπορούν να ισχύουν δύο διαφορετικές περιγραφές και να επισύρουν και διαφορετικές συνέπειες για την ίδια πράξη. Και αυτό έχει μια εξήγηση διότι τα συμφέροντα, τα διακυβευόμενα είναι διαφορετικά, άρα χρειάζεται διαφορετική προστασία και εναρμονισμένη θα έλεγα, δεν διαφέρει σε κάθε χώρα, σε κάθε χώρα ισχύει. Ξέρω τι συμβαίνει στην Ιταλία, την ξέρω πολύ καλά. Σε κάθε χώρα, λόγω υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσει, που θέλουμε και αυτή να λησαγωνοποιηθεί όπως λέμε, πρέπει να προβλέπει κάθε χώρα λοιπόν στο εθνικό της ποινικό δίκαιο το αδίκημα Τη απάτη που βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες λοιπόν, στο ποινικό δίκαιο της Ιταλίας, έχουμε το παραδοσιακό παλαιό αδίκημα έγκλημα τη Απάτη και έχουμε το αδίκημα ε, το 640α, σύμφωνα το άρθρο 640α, αδίκημα που στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ε, κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τίποτα επαναστατικό. Είναι κάτι απολύτως δίκαιο και σωστό, διότι τα διακυβευόμενα συμφέροντα είναι διαφορετικά και τα συμφέροντα είναι ευρωπαϊκά. Και αν είναι ευρωπαϊκά, όχι ταυτόσημα, χρειαζόμαστε λοιπόν μια ομοιογενοποιημένη, ε, προστασία. Σας λέω κάτι που γνωρίζετε τώρα ως πολιτικοί. Ας είμαστε πολιτικός ορθοί. Ίσως να γίνει απόπειρα σε κάποια κράτη-μέλη. Υπάρχει τάση στην κοινή γνώμη κάποιου κρατών μελών που να λέει «Ε, ευρωπαϊκά χρήματα είναι τώρα. Ακόμα και αν υπάρξει κατάχρηση δεν είναι και μεγάλο το πρόβλημα. Οπότε η προστασία των ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να είναι ευρωπαϊκό θέμα. Δεν πρέπει να αφήνεται σε ε, εθνική προθυμία του ΣΥΠΗΝ, διότι δεν υπάρχει διαπροθυμία σε όλα τα Κατημέλη για την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Ευχαριστώ. Ζήτησε το λόγο κάποιος από την αίθουσα. Κυρία μου, σας παρακαλώ, αν μπορείτε να μας, να μας συστηθείτε και να υποβάλλετε και το ερώτημά σας. ευχαριστώ πολύ που μου δίνει την ατότητα να, να μιλήσω. Στέλλα Βελίκη, φυσικός και ασχολούμαι με την πληροφορική Ευρωπαία πολίτης και με ενδιαφέρει πολύ αυτή η διάσκεψη. Ξέρω εξ ονόματος την Όλαφ και από βιβλία. Είναι πιο πολύ, έχει πολιτική χρειά περισσότερο παρά αποτελεσματικότητα. Το να δημιουργήσουμε ένα Ευρωπαίο εισαγγελέα για μένα ε, εισαγγελέα με κάνει να αισθάνομαι ότι χάνω κάποια εθνική ε, κυριαρχία. Υπάρχει ένας ε, εισαγγελέα πάνω από του εθνικού εισαγγελεί και αποφασίζει και αυτό με φοβίζει εμένα. Νομίζω ότι ήδη υπάρχει η Όλαφ. Έχει εμπειρία η Όλαφ στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Υπάρχει και ένα άτομο σε κάθε χώρα που έρχεται σε επαφή με τα θεσμικά όργανα και καταπολεμά τη διαφθορά. Υπάρχουν θεσμοί εντός των χωρών. Μιλώ για τις πριν κομμουνιστικές χώρες περισσότερο. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί που καταπολεμούν τη διαφθορά. Υπάρχει ένα άτομο της Όλαφ που μπορεί να συζητεί ή να συμμετέχει σε όλες τις έρευνες. Ε, θα μπορεί να υπάρχει καλύτερη δυνατότητα για την Όλαφ να συνεργάζεται με την Ίντερπολ. με τις αστυνομικές δυνάμεις, τις αστυνομικές υπηρεσίες που κάνουν την έρευνα. Το να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκή εισαγγελική ε, υπηρεσία ε, με νέους υπαλλήλους που θα ξέρουν τι τους ε, γίνεται, περί πρόκειται. Ένα παράδειγμα. Στις πρώην κομμουνιστικές χώρες πάντα οι ίδιοι άνθρωποι είναι πίσω από τις ίδιες εταιρείες ή έχουμε και καινούριες εταιρείες που έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά χρήματα. Είναι σαφές. Και μπορεί με τις εθνικές υπηρεσίες καταπολέμησης διαφθοράς η Όλαφ να ε, καταπολεμήσει αυτές τις εταιρείες οι οποίες ε, παρανόμως χρησιμοποιούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όταν ολοκληρώσουμε και το δεύτερο τμήμα της δημόσιας ακρόσης θα μπορέσουμε να δώσουμε μια απάντηση και στην ερώτηση αυτή. Ας περάσουμε λοιπόν στο δεύτερο τμήμα της δημόσιας ακρόασης, δίνοντας το λόγο στον κύριο Ζανό Μις, που είναι ο πρώτος Γενικός Αγγελέας του Λουξεμβούργου, και κατόπιν στον κύριο Χόρχε Εσπίνα Ράμος, που είναι εισαγγελέας από την Ισπανία Πριν όμως δώσω το λόγο στον κύριο Νίση, η κυρία Μιτερμάιερ ε, ίσως θα έπρεπε να λάβει το λόγο γιατί κάποιες ερωτήσεις είχαν απευθυνθεί και σε εκείνη. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε κάποιες από τις σημαντικές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Υπηρεσία, να διευκρινίσω τη θέση μας για αυτή τη σημαντική ευπρόσδεκτη για μας εξέλιξη. Όταν εξετάσαμε την κατάσταση και την αξιολογήσαμε όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργία Ευρωπαϊκή Εγγελική Υπηρεσία, θεωρήσαμε ότι ήταν χρυσή ευκαιρία αυτή πραγματικά για να ενισχύσουμε την επιβολή των νόμων κατά πολέμηση διαφθοράς και των απατών και του κανονισμού. Όχι μόνο σε επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Συμβουλίου τη Ευρώπη και σε άλλου διεθνεί φορεί, όπω ανέφερε ο κ. Ντένι Ντε Είμαστε πεπισμένοι ότι ο αριθμός των υποθέσεων διαφθοράς και απάτης στα, εσωτερικά, στα εθνικά δικαστήρια θα αυξηθεί αν οι έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που διεξάγεται από την Όλαφ ακολουθούνται από, παρακολουθούνται από έναν Ευρωπαίο εισαγγελέα. Ε, γι' αυτό υποστηρίζουμε τη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Εγγελική Υπηρεσία. Όσον αφορά ανησυχίε που εξέφρασε η κυρία Προλίγου, εμεί πιστεύουμε ότι παρόντο διασυνοριακή απάτη και διαφθορά και οι έρευνε για αυτά τα γεγονότα δεν γίνονται σωστά αρκετά ενεργά και δεσμεύονται οι ελεκτικές αρχές των κρατών μελών λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα των υποθέσεων, κάποιων υποθέσεων και γι' αυτό διστάζουν, είναι αργοί ή παρεμποδίζονται στην εξυχνίαση τέτοιων περιπλόκων περιπτώσεων και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό επίπεδο. Συνεπώς, οι δυνατότητες εγκαίρων καταδικών ε, είναι λίγες, περιορισμένες, αν μόνο οι εθνικές εισαγγελικές αρχές είναι υπεύθυνε. Για μας ο κρίκος που λείπει από τη διαδικασία είναι αποτελεσματική υπηρεσία ευρωπαϊκή εισαγγελία που έχει κύρος, έχει ε, τη δυνατότητα να κινηθεί για αυτές τις υποθέσεις και το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να τα αναμίξουμε αυτά με εθνικές υποθέσεις διότι τότε θα υπάρχουν διαμάχες. Αν οι αρμοδιότητες όμως είναι σαφείς, τότε ο συνδυασμός είναι καλός. Δηλαδή όλοι μπορούν να ωφεληθούν και οι αρχές που έχουμε υπόψη μας θα έχουν στο σκοπό να συντονίζουν των παραδοσιακών θεσμικών φορέων σε εθνικό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Αρχών, παραδείγματο χάρη, όπω το Eurojust και η Όλαφ είναι οι αρμόδια Ευρωπαϊκή φορεί. Μακροπρόθεσμα και από τη στιγμή θα δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Υπηρεσία, θα πρέπει να έχει σαφή εντολή που θα συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τα εγκλήματα που επηρεάζουν άμεσα τα οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σοβαρά διασυνοριακά εγκλήματα όπω διασυνοριακή διαφθορά, απάτε και άλλε πράξει. Και ίσω εδώ παντώ στον κύριο Γκάιερ. Αυτά λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, Εισαγγελική Υπηρεσία. Θα εξακολουθούμε να επεξεργαζόμεθα το θέμα και θα συνεχίσουμε και τις αποτιμήσεις μα όσον αφορά τις σχέσεις που θα υπάρχουν με διεθνείς συμβάσεις και κανόνες που ισχύουν και υφίστανται και θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στο μέλλον. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε χρόνια και χρόνια μπροστά μας για να συζητήσουμε το θέμα και είμαστε έτοιμοι. Δεύτερον, να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε για την ιστοσελίδα ε, που θα δημοσιεύει τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών πόρων. Συμφωνώ κυρία Γκρέσλε, αυτό που έχουμε για την ώρα ε, είναι ολόκληρα νεκροταφεία πληροφοριών στην Ευρώπη διότι κάθε κράτος μέλος ε, έχει δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τους δικαιούχους πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κάποιες χώρες το πραγματοποιούν πάρα πολύ καλά, δεν θέλω να υπονομεύσουμε τις προσπάθειες, τις οποίες εκτιμούμε. Το πρόβλημα είναι οι χώρες εκείνες όπου δεν παίρνουν τα πράγματα πολύ σοβαρά, δεν ενημερώνουν τις πληροφορίες και οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε μια γλώσσα που είναι δύσκολο να μεταφραστεί διότι δεν έχουν όλες οι ιστοσελίδες στα αγγλικά μεταφρασμένες πληροφορίες. Στο ερώτημά σας λοιπόν, τι θα πρέπει να συμβεί. Είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιληφθεί και θα δημιουργήσει έτσι μια πλήρη ενιαία ε, ιστοσελίδα συνοψής πληροφορίες, είτε θα το πρέπει να το κάνει η κοινωνία των ε, πολιτών. Εάν πρέπει να το κάνει αυτό η κοινωνία των πολιτών, χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις. Και η κοινωνία των πολιτών χρειάζεται να δωρητή ούτω ώστε στι τις πληροφορίες να μεταφραστούν και να συνοψιστούν. Χρειαζόμαστε πάρα πολλού ανθρώπινους πόρους στην κοινωνία των πολιτών. Πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Και μάλιστα κάνουμε σύγκριση με το τι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει ε, έχοντας τις πληροφορίες. Συμφωνώ. Ήτανε μακρά η συζήτηση επ' αυτού. Κολλήσαμε κάπου και ελπίζω ότι θα αναζωογονηθεί η συζήτηση. Και τέλος, στο ερώτημα του κυρίου Σκυλακάκη, συγγνώμη αν δεν προφέρω καλά το όνομά σας, για το βαρόμετρο, η, διαφα... η Transparency International δημοσιεύει κάθε χρόνο ε, ένα διεθνές βαρόμετρο που κάνουμε μια βολιδοσκόπηση των απλών πολιτών. Τους ρωτάμε διάφορα πράγματα, όπως δροδοκίσατε κάποιον τελευταία 12, 12 μήνες, ποιο Πιστεύετε ότι η κυβέρνησή σα είναι καλά εξοπλισμένη να καταπολεμήσει τη διαφθορά, είναι έτοιμη να κάνει κάτι τέτοιο κλπ. Και, Και είναι συγκλονιστικά τα αποτελέσματα. Οι περισσότεροι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που μα μίλησαν είπαν ότι δεν είναι πεπισμένοι ότι οι κυβερνήσει του είναι πραγματικά προετοιμασμένε να καταπολεμήσουν τη διαφθορά και την απάτη. Και όσον αφορά του περιφερειακού θεσμού, ήδη σε επικρίσει ακούστηκαν. Αυτό θα πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά και να αποκαταστήσουμε την ε, εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς όσον αφορά την καταπολέμηση της δευθοράς και της απάτης και κυρίως σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς πόρους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Μάιερ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ζανό Νις, που είναι ο πρώτος Γενικός Εισαγγελέας του Λουξεμβούργου. Ευχαριστώ. Μου είπα να μιλήσω στα αγγλικά. Δεν προτίμασα λοιπόν την παρέμβασή μου, δηλαδή την επίσημη γλώσσα της χώρας μου που είναι τα γαλλικά ή τα λουξεμβουργιανά αναγνωρίζονται. Θα μιλήσω αγγλικά και θα κάνω ό,τι μπορώ. Μου είπαν το Σάββατο ότι θα πρέπει να είναι τα λόγια του του νομικού είναι το PowerPoint, του δεν ετοίμασα λοιπόν PowerPoint. Μου είπαν ότι θα έλεγε σε πέντε λεπτά η υποτίθεται η συνεδρίαση, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι μάλλον γρήγορος. Έχω την τιμή να σας μιλήσω για τις τρεις πρωτοβουλίες που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ και 1,5 χρόνο κάποιες από αυτές, δεν είναι κάτι καινούριο. Και ξεκίνησε ήδη η δουλειά και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα άρθρα που διάβασα από την άποψη του Λουξεμβούργου, μπορώ να εκφράσω ιδιωτική άποψη, δεν μπορώ να μιλήσω σαν ε, γενικό Αγγελέας ε, ε, του Λουξεμβούργου και μέλο τη επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μπορώ να μιλήσω σαν ιδιώτη. Για την πρώτη πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το προστασία, την προστασία PIF, όπω αποκαλείται στα γαλλικά, κατά των χρήματων τη Ευρωπαϊκή Ενώσης πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποια κενά, υπάρχουν κενά. Εν συντομία θα ήθελα να αναφέρω δύο πτυχές όσον αφορά το πρόβλημα του εθνικού ουσιαστικού δίκαιου και για την αμοιβαία νομική συνδρομή. Και αυτά πάλι από την πλευρά του Λουξεμβούργου. Με τα χαρά σας λέγω κάτι που δεν θα σας εκπλήσει ότι η χώρα μας είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε ποινικοποίησει και ενσωματώσει στο εθνικό μας δίκαιο όλες τις συμβάσεις PIF με αυστηρές πίνες φυλάκισης από ένα μήνα μέχρι πέντε χρόνια και μπορεί μέχρι δέκα χρόνια η κάθριξη σε κάποιες περιπτώσεις σύμφωνα με κάποιους νόμους και πρόστιμα μέχρι 30.000 ευρώ μπορούν να επιβληθούν χωρί να λησμονούμε και κατάσχεση και αποκατάσταση πόρων και ανάκτηση πόρων που είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό σε κάποιε περιπτώσει από ότι είναι το πρόστιμο που επιβάλλεται. Το σημαντικότερο επίσης ότι είναι, ε, παρομοιάζεται με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος το δίκημα αυτό κατά της, των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Επίσης λοιπόν και αυτός που χρησιμοποιεί τα χρήματα ε, τιμωρείται και αυτός που έκανε την κλοπή. Λοιπόν, να σας πω γιατί σας λέω αυτά τα πράγματα, για να σας πω ότι από τη δική μας άποψη και πρόσθετη ποινικοποίηση δεν θα δώσει προστιθέμενη αξία όχι μόνο από την άποψη την εθνική αλλά και τη διεθνή διότι μέχρι τώρα δεν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα όσον αφορά και την αμοιβαία νομική ε, αρρωγή όσον αφορά την ε, περιπτώσει αυτές καταπολέμηση των απατών κατά των, κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Λοιπόν, η αμοιβαία νομική αρρωγή και σχετική πρωτοβουλία όσον αφορά τη σύμβαση PIF, πρέπει να σας πω ότι είχαμε προβλήματα κάποιες φορές, αλλά δεν ήταν νομικής φύσεως. Και είχα την ευκαιρία να μιλήσω στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών πριν από δύο χρόνια και το ίδιο είπα και τότε όπως και τώρα. Αν έχουμε προβλήματα σε 99% των υποθέσεων, τα προβλήματα είναι συνήθως πρακτικής φύσεως κάποια ανόητα πρακτικά προβλήματα. Δεν μιλάμε μια κοινή γλώσσα. Η μετάφραση από γλώσσα χ προς αγγλικά και γαλλικά ε, δεν είναι βανάγνωστη. Δεν μπορώ να βρω έναν αριθμό τηλεφώνου. Αυτά είναι πρακτικά προβλήματα. Δεν είναι νομικά προβλήματα ανεπίλητα ε, που μπορούν να επιληθούν από νέες νομοθεσίες, αλλά μέσω πρακτικής προσέγγισης. Και εκτιμώ πολύ το έργο του Eurojust, και το, του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για τα ποινικά θέματα. Στο κείμενο που δημοσιεύθηκε περιγράφουμε την κατάσταση στο Λουξεμβούργο. Μπορείτε όλοι να διαβάσετε. Δεν θα σας διαβάσω το κείμενο, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Απλουστεύω. Μπορούμε να απαντήσουμε σε τι μας υποβάλλονται ως χώρα όσον αφορά τα θέματα ε, καταπολεμήσεως των απατών αυτών. Να σας διευκρινίσω κάτι που αφορά εσάς περισσότερο. 400, με 400 αιτήσει δεχόμαστε κάθε χρόνο. Για αμοιβαία Και βλέπουμε ότι αυτοί πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα ε, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τα νέα κείμενα που θεσπίζονται και τα ποικίλα κείμενα. Αντί να υπάρχει ένα κείμενο για την αμοιβαία ρογή, οι νομοθέτε εσείς δημιουργείτε όλο και περισσότερου νόμους και κείμενα και είναι πολύ δύσκολο αυτοί πρέπει να εφαρμόσουν τους νόμους να βγάλουν άκρη με όλα αυτά τα κείμενα. Και θυμάμαι πολύ καλά όταν ε, παρουσ... Λοιπόν, διαβάσαμε σε μια υπόθεση ότι στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα μοναδικό ενιοποιημένο κείμενο. Και συζητείται ακόμα σήμερα η πρόταση και πόρα που έχουμε από ένα ενοποιημένο κείμενο. Και εμείς οι δικαστές δεν είμαστε όλοι δικευμένοι. Σε μικρή περιφέρεια, μικρό νομό, μικρό, μικρή επαρχία μπορεί ο δικαστής να έχει μία-δύο υποθέσεις ε, το χρόνο και δεν μπορεί να βγάλει άκρη και πάλι. Σας συστήνω, να κρατήσουμε τα πράγματα απλά. Εάν μπορούσαμε να κινηθούμε με ένα κείμενο, κινηθούμε με ένα κείμενο. Πολλά υπόθηκαν για την Όλαφ ήδη. Κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Και συμφωνώ με τον Διευθυντή Κέσλερ. Υπάρχουν αρκετά εκρεμή θέματα και σε εθνικό επίπεδο. Και λένε οι δικαστές, τι αξίζει αυτό που μου λένε, είναι μάρτυρες αυτοί, είναι πυρογνώμονες. Τι γίνεται αν ε, ε, Επίση συμμετέχει στην υπόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρείται εμπειρογνώμονη ή όχι. Αυτά είναι το έθεσε η Δόκτωρ Κέτλερ. Νομίζω ότι χρειάζεται νέα διευκρίνηση και ίσως νομοθεσία για το ίδιο θέμα, η Eurojust. Το Eurojust ακόμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά και δεν έχει εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εμείς στο Λουξεμβούργο επανειλημμένως ε, μπορούμε, το έχουμε κάνει, μπορούμε να πάμε στη Χάγη, το κάναμε, συνεργαζόμαστε άριστα με τους εκπροσώπους μας εκεί. Όμως, δεν πρέπει να κάνουμε αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξουσία κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας να ξεκινούν ποινικέ έρευνες. Γιατί? διότι τώρα έχουν πλήρη εμπιστοσύνη από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για διευκόλυνση, για βοήθεια, για μεσολάβηση μεταξύ διαφόρων εθνικών διοκτικών αρχών και θεωρούνται σαν ουδέτερος φορέας. Και αυτή η θετική πτυχή δεν θα πρέπει να υπονομευθεί δίνοντάς τους εξουσίες όπως συζητήθηκε ήδη σήμερα, να τους δώσουμε την εξουσία να επιβάλλουν την άποψή τους επιθυνικών διοκτικών αρχών. Δεν είναι εκεί για αυτό το σκοπό. Πολύ καλά κινούνται σήμερα και έτσι πρέπει να παραμείνει η κατάσταση. Και κάτι συζητήθηκε και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Δεν θα πρέπει να βγει εκτός Eurojust. Η Eurojust θα πρέπει να παίξει το ρόλο που παίζει που είναι θετικότατος και δεν χρειαζόμαστε άλλη εισαγγελική αρχή. Ο Δόκτωρ Κέσλερ αναφέρθηκε στο πώς θα έπρεπε να συσταθεί. Αποκεντρωμένη υπηρεσία εισαγγελική ευρωπαϊκή που είναι μάλλον μια φικτή λύση και δεν συμφωνώ μαζί σας ότι είναι κατά η εθνική Όλο και περισσότερο είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Αγγελική Υπηρεσίας από τη στιγμή που θα συσταθεί με τέτοιο τρόπο που θα σέβεται τις εθνικές ιδιοξυγκρασίε ιδιαιτερότητε. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Όπως και ε, οι όλοι οι δικαστές εθνικοί είναι για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ε, εθνικοί δικαστέ πρωτοδικίου. Πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικό ρόλο. και θα πρέπει να, η υπηρεσία αυτή να είναι κοντά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ενδεχομένω στο Λουξεμβούργο. Αυτό είναι κάτι πολιτικό που θα πρέπει να επιληθεί αλλού και θα το συζητήσω εγώ. Που θα δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Συρρεπία, Υπηρεσία. Τώρα η πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ξέρουμε ότι η διαφθορά δεν γίνεται αντιληπτή προφανώς σαν ποινική συμπεριφορά από όλου. Ξέρουμε ότι είναι, ξέρουμε πόσο κοστίζει στις οικονομίες, και ότι υπάρχει η διαφθορά. Διάβασα ότι αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μία έκθεση για καταπολέμηση διαφθοράς κατά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ναι, αλλά προσοχή, υπάρχουν κάποια μικρά κράτη-μέλη και ξέρω από κάποιον, κάποιος από εσά που μιλά, είναι σε όλες επιτροπές αξιολόγησης. ΟΣΑ, ΦΑΤΦ, Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πολλές επιτροπές αξιολόγησης συμμετέχω και συμβαίνουν πολλά κάθε χρόνο σε αυτό το θέμα. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος, ε, μεγάλος φόρτος εργασίας και συνεχώς οι συνάδελφοί μου και εγώ επενδύουμε χρόνο στην αξιολόγηση, αυτός ο χρόνος χάνεται από αποτελεσματική δουλειά. Εντάξει, είναι σημαντική αξιολόγηση και βλέπουμε και εμείς πράγματα τα οποία δεν ξέραμε. Είναι κάτι σημαντικό αλλά δεν θα πρέπει να αυξηθεί υπερβολικά φόρτος εργασίας. Κάτι που δεν συζητηθήκε ακόμα σήμερα. Οι διάφορες μονάδες ε, καταπολεμήσεως του οικονομικού εγκλήματος είναι σημαντικές. Το περασμένο Σάββατο έγινε μια διάσκεψη στο Παρίσι του FETF όπου εκεί συμμετέχουν διάφορε ομάδε κατά πολεμήσεω τη διαφθορά και παρουσιάστηκαν δύο σημαντικά έγγραφα στη διάσκεψη. Πρώτα απ' όλα, ευέλτιστε πρακτικέ για τη χρήση των συστάσεων ΕΦΕΤ για την καταπολέμηση τη διαφθορά. Υιοθετήθηκε στη διάσκεψη. Εμπεριέχει σημαντικότατε ιδέε για το πώ οι μονάδε εξυχνίαση οικονομικού εγκλήματο μπορούν να συμμετάσχουν στη μάχη και ομάδα έγματ λευκή βίβλος για το ρόλο που μπορεί να παίξει διάφοροι φορεί στην εξυχνίαση των οικονομικών εγκλημάτων και την ανάκτηση ε, των πόρων. Αυτό έχει τεράστια υπεραξία το έγγραφο. Γιατί? Διότι Η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών συλλέγει πληροφορία από τη στιγμή που η διαφθορά είναι σε οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή, αν εγώ πάρω ένα ρόλεξ το οποίο είναι παραποιημένο, δεν θα το δει κανεί. Αλλά ε, θα διαπιστωθεί αν υπάρχει η διαφθορά, έχει διαπραχθεί με χρήματα. Καλό εσάς σαν νομοθέτες να κάνετε αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματική εποπτεία της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, ομάδων συμφερόντων, να υπάρχει ελευθεροτυπία. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό οι νομοθέτες να έχουν αρκετό θάρρος για να επιβάλλουν αυστηρέ ποινικέ ε, κυρώσει και να καθαρίσουν πρώτα τα του οίκου του απαλλασσόμενοι από ιεσδήποτε ασυλίες που καμιά φορά είναι εκεί για να προστατεύουν τους ίδιους. Αυτά λοιπόν, αυτά θα σας πω σήμερα. Μπορείτε να διαβάσετε τα υπόλοιπα στο έγγραφό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και προσβλέπω στη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε κύριε Ζανοτνιές. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ε, Χόρχε Σπίνα Ράμος που θα μας ε, κάνει μια παρουσίαση εκ μέρους ε, της ε, Ισπανικής Γενικής Εισαγγελίας με θέμα και πάλι τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πάταξη της απάτης και της διαφθοράς. Κύριε Σπίνα, έχετε το λόγο. Thank uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και προσωπική αλλά και εκ μέρους ε, του Ισπανικού, Ισπανού Γενικού Εισαγγελέα να σας παρουσιάσω την γνώμη μας για το θέμα αυτό και την εμπειρία που έχουμε από θέματα όπως αυτό που εξετάζουμε σήμερα. Μου είπε να μιλήσω στα αγγλικά, γι' αυτό και δεν θα μιλήσω στα ισπανικά. Επίσης μου είπαν να κάνω την παρουσίαση μου με PowerPoint. Όπερ και γένετο, γιατί ως εισαγγελέα και πειθαρχημένος άνθρωπος έφερα το PowerPoint μου και στα αγγλικά και μου είπαν ότι θα συμπεριληφθεί και στην ιστοσελίδα σας μια και δεν έχετε προλάβει να λάβετε την παρουσίασή μου μέχρι τώρα. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω συντομία τι κάνουμε εμείς ό,τι αφορά τα δικήματα που εμπίπτουν στη σύμβαση PIF, στη Σύμβαση για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και θα επικεντρωθώ σε αυτό που κάνει η Ισπανία, γιατί κατά τη γνώμη μα δεν μπορούμε να μιλάμε ε, για εγκλήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων τη Ένωση μόνο υπό το εθνικό πρίσμα. Θα πρέπει να έχουμε μια και πιο γενική πανευρωπαϊκή προσέγγιση, γιατί αυτή η προσέγγιση απαιτείται για να καταπολεμηθούν τέτοιου είδου διασυνοριακά εγκλήματα. Έχουμε αρκετές ε, εγχώριες πρωτοβουλίες, δεν πρόκειται να τις αναλύσω διεξοδικά. Έχουμε πολλές εθνικές πρωτοβουλίες προκειμένου να βελτιώσουμε το σύστημά μας και τις δικανικές δομές και τις διοκτικές δομές μας, ε, λαμβάνοντας υπόψη το δίκαιο και το ουσιώδες ποινικό δίκαιο και το δικονομικό ποινικό δίκαιο, ε, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και το κοινοτικό δίκαιο, υιοθετώντα μια διπλή προσέγγιση για να οδηγηθούμε σε πιο επιτυχή αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις που είχαμε στην Ισπανική Εισαγγελική Αρχή, θα ήθελα να πω ότι ε, έχουμε εργαστεί εργοδός προκειμένου να βελτιώσουμε την εξειδίκευση των επιμέρους εγγελέων και μάλιστα προσπαθήσαμε να αφυπνίσουμε όλους τους εισαγγελεί για το τι σημαίνει ο ΛΑΦ, τι κάνει ο ΛΑΦ, τι σημαίνει η πράσπιση των οικονομικών συμφερόντων, να μην θεωρηθούν αυτά ως δεδομένα, γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί δικαστές, τόσοι πολλοί εισαγγελεί που δεν έχουν ιδέα για το τι είναι η ΟΛΑΦ και τι κάνει η ΟΛΑΦ, ποιο είναι το έργο της ΟΛΑΦ. Γι' αυτό και κρίναμε σκόπιμο να βελτιώσουμε την κατάρτιση και την ενημέρωση των εισαγγελών και από διαρθρωτική άποψη, και από θεσμική λοιπόν, θα ήθελα να σας πω τι κάνουμε σε ό,τι αφορά την πάταξη της διαφθοράς. Είναι σημαντικό να το δούμε και υπό το κοινοτικό πρίσμα. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεννόησης και συνεργασίας με την ΟΛΑΦ ήδη από το 2008, κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα προκειμένου να δεχθούμε τα αποδεικτικά στοιχεία και το ερευνητικό υλικό που μας έχει ε, κοινοποιήσει η ΟΛΑΦ σε διάφορες ε, δίκες. Απλώς χρησιμοποίησαμε τον κανονισμό 1073, άρθρο 9 συγκεκριμένα, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ε, δώσαμε τη δυνατότητα στην ΟΛΑΦ να λάβει μέρος στη δίκη ως πολιτική αγωγή. Εν συντομία, Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η βασική μας διάρθρωση για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς σε επίπεδο εισαγγελία. Έχουμε ένα ειδικευμένο γραφείο δίωξης της απάτης με 16 ε, εισαγγελείς και αντισαγγελείς σε διάφορα μέρη της Ισπανίας. Η μεγαλύτερη διαφορά, αν το συγκρίνουμε με άλλες αγγελικές αρχές, είναι ότι εμείς έχουμε και κάποιες ε, άλλες μονάδες στις οποίες συμμετέχουν ελεκτές και ένα φορολογικό γραφείο. Έτσι έχουμε ένα πολυτομεακό περιβάλλον, πολυσχηδές και μπορούμε να, να διερευνήσουμε πολύ πιο περίπλοκες περιπτώσεις. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αρκεί μια μηγής νομική γνώση που κατέχει ο εισαγγελέας, αλλά χρειάζεται η συνδρομή και άλλων ειδικευμένων όπως είναι ελεγχτές, φορο, εφοριακοί κτλ. Επίσης έχουμε αυτή την περιφερειακή διάρθρωση, 16 εισαγγελείς στις α, ε, αυτόνομες περιοχές, αλλά έχουμε και ε, αντιπροσώπους των εισαγγελέων που ορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και ανάλογα με τον αριθμό των υποθέσεων που έχουμε. Γιατί το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά σε ορισμένε περιφέρειε εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα. Αυτοί λοιπόν οι αντιπρόσωποι του εισαγγελέα έχουν διπλή ιδιότητα είναι τοπική Ε, εμπίπτουν στα κεντρικά γραφεία της Σεβίλης, Μάλαγα, Βαρκελόνης, αλλά ταυτόχρονα εμπίπτουν ε, και καλύπτονται από τη, από τη Γενική Εισαγγελία Δίωξης ε, του Οικονομικού Εγκλήματος. Φυσικά αντιμετωπίζουμε προβλήματα, δεν μπορούμε να πούμε ότι μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε είμαστε απολύτω ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα. Αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα στην πράξη και συμφωνώ με τον συνάδελφο από το Λουξεμβούργο ότι τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι νομικού χαρακτήρα, αλλά πρακτική υφή. Δηλαδή θα θέλαμε πολύ πιο αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Δυστυχώ δεν υπάρχουν τέτοια αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των διαφόρων υποθέσεων, δεν μας βοηθάει και πολύ στο γεγονό ότι το ισπανικό σύστημα στηρίζεται σε μεμονωμένους ανακριτές δικαστές, σε ατομικές, ατομικούς ε, και η γίνεται γενική καθοδήγηση από τον εισαγγελέα, μπορεί να γίνει και το αντίστροφο. Μπορεί συχνά ένα εισαγγελέα να συνεργάζεται με έναν ανακριτή ή διοικητικό δικαστή. Κάτι που καθιστά πολύ δύσκολη την παρακολούθηση τέτοιων υποθέσεων. Τώρα, αν μιλούμε μόνο υπό το πρίσμα του γραφείου του εισαγγελέα, είναι πολύ δύσκολο ε, να ενημερώνει 2.000 και εισαγγελείς που δεν είναι ειδικευμένοι για τέτοιου ε, εγκλήματα, να τους ευαισθητοποιήσω ότι αφορά την ανάγκη συχνής ενημέρωσης ε, και αναφοράς προκειμένου να παρακολουθούνται οι υποθέσεις. Επίσης αντιμετωπίσαμε προβλήματα και σε ό,τι αφορά το στενό χρονικό περιθώριο από την ε, ενημέρωση της ΟΛΑΦ υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις και κολλησιεργίες και σε εθνικό επίπεδο, όχι μόνο σε περιπτώσεις της σύμβασης ΠΙΦ, της ε, Σύμβασης Προστασίας των Οικονομικών Συμφερόντων της Ένωσης, αλλά πολλές φορές ε, οι διοικητικές έρευνες που ξεκινάει ο ΛΑΦ χρησιμοποιούνται ως ε, σύστημα έγκυρης προειδοποίησης για κάποιους υπόπτους Ε, που λαμβάνουν τότε τα μέτρα τους, κάτι που καθιστά πιο δύσκολη αργότερα την ποινική δίωξη, την ανάκριση, γιατί είναι δύσκολη η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, μια και στο μεταξύ έχουν ψηλιαστεί την κατάσταση από την έναρξη των διοικητικών ερευνών της ΟΛΑΦ. Τώρα, Πιστεύω ότι πέραν των εθνικών προσπαθειών και δομών χρειαζόμαστε συνεργασία και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε την ε, αναθεώρηση της ΟΛΑΦ, έχουμε τη σύμβαση ΠΙΦ, Έχουμε και τη Eurojust που είναι ένα συντονιστικό, ένα συντονιστικός φορέας, το αναφέρατε και αυτό. Οπότε μπορούμε επιτέλους να υλοποιήσουμε αυτή την ιδέα ότι τα σύνορα που εξαφανίστηκαν για τους ε, πολίτες και για τους εγκληματίες δυστυχώς εξακολουθούν να ορθώνονται για τις ε, αστυνομίε και τους δικαστικούς και εισαγγελίες. Επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τα νέα εργαλεία που προτείνονται. Για παράδειγμα, το πακέτο πάταξης της διαφθοράς που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι, την μεταρρύθμιση της ΟΛΑΦ που ακούσαμε σήμερα, τη δυνατότητα χρήσης του ποινικού δικαίου με τον τρόπο που πρότεινε πρόσφατα στην ανακοίνωσή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η λισαβονοποίηση, η ένταξη δηλαδή της σύμβασης PIF στη συνθήκη της Λισαβόνας. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ σωστά βήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Επίσης η ενίσχυση της Eurojust, της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας και εκεί υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις, γιατί η απόφαση δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως από όλα τα κράτη-μέλη και υπάρχουν οι νέε δυνατότητε που μα δίνει το άρθρο 85 τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, εσεί θα αποφασίσετε αν εκεί υπάρχουν κάποιε βελτιώσει που είναι σκόπιμο να γίνουν ή κάποιε περαιτέρω ρυθμίσει στο μέλλον. Πάντω, για του νέου μηχανισμού και τα νέα εργαλεία, προσπαθώ να ολοκληρώσω, και πάλι έχουμε την πρόταση ΕΠΟ της Ευρωπαϊκής Αγγελική Αρχή αυτή η πρόταση είναι πολύ διορατική και προχωρημένη στην προσπάθεια καταπολέμησης των αδικημάτων που εμπίπτουν στην σύμβαση ΠΙΦ, της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων. Εμείς μελετήσαμε την κατάσταση και, και την πρόταση και θεωρούμε ότι πραγματικά ε, περιέχει μια προστιθέμενη αξία. Γιατί μας βοηθάει όχι μόνο να εργαστούμε καλύτερα και κάπως διαφορετικά σε σχέση με τις δυνατότητες που μας δίνουν οι προηγούμενοι μηχανισμοί. Πραγματικά έμεινα εμβρόντιτος από την άποψη ενός συναδέλφου ότι η Εθνική Εισαγγελία είναι κατά τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Αγγελική Αρχή. Εγώ την αντίθετη αίσθηση έχω. Το αντίθετο πιστεύω ότι ούτω ή άλλω ε, στο συμβουλευτικό φόρουμ των Γενικών Εισαγγελέων, οι εισαγγελίε ούτω ή άλλω ε, συνέρχονται δύο φορέ το χρόνο και μερικέ φορέ και περισσότερε φορέ ε, και συζητούν και οι εντυπώσει που έχω αποκομίσει από τι συναντήσει αυτέ είναι αντίθετο ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη τη πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Μπορεί τα κράτη-μέλη να μην έχουν λάβει ακόμη την απόφαση σχετικά. Πάντως η δημόσια κατηγορία, η εθνική εισαγγελείς έχω την αίσθηση ότι είναι υπέρ της πρότασης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Και τώρα να αναφερθώ σε ένα πιθανό μοντέλο που είναι το μοντέλο που κρίνουμε εμείς ως το καλύτερο από άποψη κόστος κόστος-οφέλους αλλά και από το πρίσμα ότι η νέα πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή δεν θα εκλειφθεί ως το νέο σώμα που θα εισβάλλει στην εθνική δικαιοδοσία. Πιστεύω ότι το μοντέλο που προτείνουμε θα αποφύγει, θα αυτό το κίνδυνο. Είναι μια μικρή κεντρική δομή με επικεφαλή στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και θα υπάρχουν αντιπρόσωποι του κατά το ισπανικό σύστημα εκπρόσωποι, το αντιπρόσωποι του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στα κράτη-μέλη, στις εθνικές δικαιοδοσίες, που θα έχουν αυτή τη διπλή ιδιότητα, αυτή η εξουσιοδοτημένη από τον Γενικό Εισαγγελέα τον Ευρωπαίο στα κράτη-μέλη, θα έχουν και τις γνώσεις και τις γλωσσικές και τις τοπικής κατάστασης και θα διευκολύνουν το έργο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Επίσης, η Eurojust θα πρέπει να συνεπάρχει με την πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Δεν θεωρούμε ότι η Eurojust θα μετατραπεί στον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Άλλο η Eurojust, άλλο... άλλες οι αρμοδιότητες και η αποστολή τη Eurojust και άλλο η αποστολή και οι του ΕΠΟ. Πιστεύουμε θα πρέπει να διατηρηθεί λοιπόν και η Eurojust. Επίσης, η ΟΛΑΦ θα πρέπει να, αποτελέ, να αποκτήσει εξουσίες ώστε να αποτελέσει μια πραγματικά οικονομική αστυνομία, μια υπηρεσία δίωξη του οικονομικού εγκλήματο, υπό την αιγίδα ίσω τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Έτσι, δεν θα έχουμε το πρόβλημα ότι μερικέ φορέ ότι η Όλαφ περιορίζεται μόνο σε διοικητικέ έρευνε και θα μπορούμε ήδη από την αρχή, με όλη την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία, την πλούσια εμπειρία που έχει συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια η ΟΛΑΦ, να ξεκινά ταυτόχρονα ποινικέ έρευνε, ανακρίσεις ε, υπό την αιγίδα φυσικά της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής, χρησιμοποιώντας όμως όλα τα εργαλεία που έχει η Όλαφ και τα νέα εργαλεία που θα της δοθούν ενδεχομένω. ο κύριος Κέσλερ μάλλον, ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ, είπε κάτι στην αρχική του ομιλία που είναι πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει να γίνει ένα ποιοτικό άλμα με τις νέες προτάσεις. Αλλιώς θα είναι σαν να βελτιώνουμε μία παλιά δομή που όσο καλή και γίνεται με τις βελτιώσεις ε, θα παραμείνει στο χαμηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας εξαιτία της παλαιότητάς της. Ενώ η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει πολύ περισσότερες ε, νέες δυνατότητες. Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ράμος. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο του Λουξεμβούργου, πρώτο γενικό εισαγγελέα, καθώς επίσης και τον κύριο Χόρχε Σπίνα Ράμος. Έρχεται τώρα η ώρα των ερωτήσεων και της συζητήσεως. Αν επιθυμεί κανείς να ερωτήσει, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Αλλιώς να δώσω το λόγο. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Πρώτα στον κύριο Γκάιερ, μετά στην κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους κυρίους Νίς και Εσπίνα. Έμαθα πολλά πράγματα και είμαι, ε, νιώθω ευχάριστη έκπληξη διότι η εικόνα που μεταφέρουν πολλοί εδώ, άλλοι, σχετικά με την στάση των εθνικών εισαγγελέων είναι πολύ διαφορετική. Αυτά δηλαδή που ακούμε στους διαδρόμους από αυτά που μας βεβαίωσαν τώρα οι δύο κύριοι. Τώρα, και από τις δύο αυτές παρεμβάσεις δεν αντελήφθη και γι' αυτό παρακαλώ να το διευκρινίσετε. Πού βλέπετε τους λόγους για το ότι είναι τόσο μικρές, τόσο περιορισμένες οι διώξει στο εθνικό επίπεδο. Γνωρίζουμε δηλαδή από τις εκθέσεις της Όλαφ ότι οι υποθέσεις που διώκονται στο εθνικό επίπεδο, που καταλήγουν δηλαδή σε απαγγελία κατηγοριών, δυστυχώς δεν είναι τόσο υψηλός αριθμό αριθμός αυτός όσο θα επιθυμούσαμε. Από τις παρεμβάσεις σας αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο κύριος Νης σε κάποιο σημείο είπε ότι είναι προβλήματα πρακτικού χαρακτήρα σε 99% των περιπτώσεων. Άρα και εδώ, και ρωτώ δηλαδή κάπως πιο προβοκατόρικα ας πούμε, έχει σχέση για παράδειγμα με το γεγονός ότι λαμβάνεται εκθέσει της Όλαφ σε γλώσσες που ενδεχομένως είναι απολύτως συμπτωματικό να έχετε κάποιον στο γραφείο σας που να μιλεί τη γλώσσα αυτή και να μπορεί να καταλάβει το ντοσιέ. Κάτι τέτοιο θα είναι πραγματικά συγκλονιστικό εάν τα προβλήματα είναι τέτοιου χαρακτήρα. Και βέβαια πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το λύσουμε αυτό. όσοι άνθρωποι που ασκείτε την πρακτική στις χώρες μέλη, δηλαδή ε, ασχολείστε στην πράξη με τα θέματα αυτά, με τις υποθέσεις που σας παραπέμπει όλα αυτά, πού βλέπετε τα προβλήματα και πώς θα θέλατε να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή στο μέλλον. Τώρα ας παίξω λίγο το συνήγορο του διαβόλου και ας καθίσω τώρα στο έδρανο του Συμβουλίου. Ας πω λοιπόν, δεν το θέλω δεν το θέλω αυτό τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα. Έχω λοιπόν δύο δυνατότητες να σταματήσω την πορεία αυτή. Πρώτο το θέμα της έδρας. Το είπε ο κύριος Νης. Ναι, εσείς προτείνατε το Λουξεμβούργο βέβαια. Άλλωστε είναι πολύ συμπαθητικό αυτό εκ μέρους σας. Εν μέρη μάλιστα χαίρετε, χαίρετε και της υποστήριξής μου. Αλλά με την μετακίνηση του Γραφείου Ευρεσιτεχνιών Μόναχο, Λονδίνο, Παρίσι ήταν τότε και οι χώρες οι οποίες μας ζητούν περικοπές και εξοικονομήσεις είναι οι χώρες όπου βρίσκεται το Μόναχο, το Παρίσι και το Λονδίνο. Δεν είναι βεβαίως ικανοποιημένοι τελικά οι χρηματοδότες που πρέπει και να εξοικονομήσουν από πάνω. Αν λοιπόν δεν θέλει το Συμβούλιο την Ευρωπαϊκή Γενική Αγγελία θα κάνει τρεις προτάσεις που δεν θα ικανοποιήσουν κανένα για την έδρα και θα μπλοκάρει το θέμα στην ουσία επάπειρον. Μετά θα τονίσει βέβαια και με ιδιαίτερη έμφαση το κόστο των μεταφράσεων και πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν τα θέλουμε εμεί αυτά τα πράγματα και γι' αυτό ευχαριστώ για το θέμα της έδρας που τονίσατε και δεν το λέω αυτό για να κάνουν αντιπολίτευση κανένα. Είναι πραγματικό το θέμα. Το δεύτερο είναι τα πρακτικά προβλήματα που ε, ε, εντοπίσατε. Αντιλαμβάνομαι ότι σας ενδιαφέρει να έχετε τις, καλύτερε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις μεταξύ εθνικών ε, εισαγγελικών αρχών και ευρωπαϊκού επίπεδου. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη, δηλαδή πώς θα λυθούν εκεί τα προβλήματα. Πού βλέπετε λοιπόν να εντοπίζονται τα προβλήματα στο επίπεδο των εθνικών εισαγγελικών αρχών για την επεξεργασία των υποθέσεων που τους ε, ε, παραπέμπει η Όλαφ, ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν, πώς θα μπορέσει να εξασφαλιστεί η ορθή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής εισαγγελία και Εθνικών και πού εντοπίζονται τα πρακτικά προβλήματα. Είναι η γλώσσα. Είναι ενδεχομένω οι εκθέσει τη Όλαφ οι οποίε κάπω δεν εντάσσονται μέσα στα δικά σας δικονομικά συστήματα. Καμιά φορά είναι απλά πράγματα τα οποία ωστόσο μπορούν να λυθούν. Ευχαριστώ κύριε Γκάιερ. Η κυρία Κρέσλε. Ευχαριστώ. Τα νούμερα για το Λουξεμβούργο. Οι υποθέσεις δηλαδή που παρέπεμψε η Όλαφ μεταξύ 2006 και 2011, δύο για το Λουξεμβούργο, για την Ισπανία 54 υποθέσεις. Τουλάχιστον στο Λουξεμβούργο υπήρξε μια καταδίκη, στην Ισπανία το ποσοστό ήταν 9,3%. Ε, δεν μου φαίνεται μεγαλειώδες. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Ισπανό εισαγγελέα πώς μπορεί να σχολιάσει. Ούτε και για το Λουξεμβούργο μου φαίνεται μεγαλειώδες. Αλλά τι να πω. Στο Λουξεμβούργο είναι και 10.000 ευρώ υπάλληλοι. Και μου φαίνεται περίεργο που να μην σημειώθηκε καμιά υπόθεση. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι στις εσωτερικές της έρευνες η Όλαφ είναι πάρα πολύ ας πούμε αυτοσυγκρατημένη σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που διοχετεύει. Αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι δεν χρειαζόμαστε καν τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα διότι έχουμε εθνικές διαδικασίες που λειτουργούν καλά. Η ιδέα για έναν εθνικό εισαγγελέα με ευρωπαϊκές αρμοδιότητες μου φαίνεται καλή, αλλά τι θα κάνουμε με τις υφιστάμενες διαρθρώσεις. Θα ήθελα από τον Ισπανό εισαγγελέα να μου πει ποια είναι η γνώμη του για τον εθνικό ευρωεισαγγελέα, στον πούμε έτσι. Μετά, στο άρθρο 86 της Συνθήκης της Λισαβόνας λέει ότι όλα αυτά ξεκινούν από την Eurojust, για την οποία δεν έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα. Ούτε η Όλαφ μιλεί για την Eurojust, σαν να μην υπάρχει. Και γι' αυτό, πώς βλέπετε τη συνεργασία με την Eurojust για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και ποια πράγματα πρέπει να βελτιωθούν. Εάν δεν λειτουργούν οι εθνικές εισαγγελικές αρχές στον τομέα αυτό, δεν θα λειτουργήσει ούτε ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας. Αυτό θεωρώ εγώ. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι πώς θα μπορέσουμε να παρακινήσουμε τις εθνικές εισαγγελικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Πέστε μας μερικές εμπιστευτικές συμβουλές, αν μπορώ να το πω έτσι. Είπατε ακόμα, ξεφορτωθείτε, είπατε, όλες τις ασυλίες. Όταν ακούει ο βουλευτής ασυλία, αμέσως σκέφτεται την κοινοβουλευτική ασυλία. Αλλά είναι και η ασυλίες των υπαλλήλων. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί, ποια είναι η βάση για το, για το έτοιμά σας αυτό. Πρώτα απ' όλα ο κ. Γενικό Συγγελέα του Λουξεμβούργου και μετά ο κ. Ράμος. Ευχαριστώ. θα μου επιτρέψετε να πατήσω στα γερμανικά στην κυρία Γκρέσλερ. Πρώτα στον κύριο Γκάιερ βέβαια. Συνεργασία λοιπόν πρώτα. Και πού εντοπίζονται τα προβλήματα στη συνεργασία με την Όλαφ. Έχουμε ορισμένα προβλήματα με την Όλαφ. Το μεγαλύτερο που είχαμε στην πράξη είναι η μακρά χρονική περίοδος πριν να γίνει η παραπομπή στην Εθνική Αρχή. Δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον ανακριτή, τον οποίο έχουμε εμείς, το θεσμό του ανακριτή, να πάει να διεξαγάγει μια έρευνα σε μια κατοικία, ας πούμε, όταν στην ουσία ήδη η Όλαφ, καμιά φορά και η Eurojust, έχουν προαναγγείλει ότι θα πάνε διότι δεν μπορεί να παρέμβει η εισαγγελική αρχή με τρόπο που να τους ευνηδιάσει. Πρέπει επίσης να γίνει μια ενιαία ρύθμιση για τα όσα διαπιστώνει η Όλαφ και πανευρωπαϊκά διότι αλλιώς υπάρχουν ατελείωτες συζητήσεις κατά πόσον τα, οι ενδείξεις της Όλαφ είναι ισχυρές παντού. Τώρα το γλωσσικό δεν αποτελεί πραγματικά πρόβλημα για το Λουξεμβούργο. Ίσως οι άλλες χώρες όμως, οι οποίες έχουν λιγότερη επαφή με ξένες γλώσσες και δεν είναι δίγλωσσες ή και τρίγλωσσες όπως είναι σε πολλές περιπτώσεις οι κάτοικοι του Λουξεμβούργου. Μπορούν να ρυθμιστούν όμω τα πράγματα αυτά, εφόσον επιθυμεί κανεί, λέει ο κ. Γκάιρ. Βεβαίω, έχετε δίκιο. Έρχομαι στην κυρία Γκρέσλε. Πώ θα κάνουμε τι αγγελικέ αρχέ να δουλέψουν. Με το κνούτο, θα, έλεγε, θα μπορούσε να πει κανεί, αλλά βέβαια δεν προσφέρει πολλά αυτό. Το περισσότερο, το καλύτερο μάλλον, είναι η ευαισθητοποίηση των δικαστικών αρχών για την ανάγκη προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ενώσεως. Αυτό γίνεται εδώ και καιρό. Είμαστε σύμφωνοι ότι πρέπει να συνεχίσει να γίνεται η προσπάθεια αυτή. Πολλές δικαιοδοσίες της περιφέρειας συνήθως συχνά λένε «Μα δεν ενδιαφέρει αυτό, είναι χρήματα των Βρυξελών». Αυτή η αντίληψη πρέπει να πάψει να υπάρχει. Στην πρωτοβουλία της Κομισιόν αναφέρεται και η ΣΕΠΟΛ. Δηλαδή η κοινή ευρωπαϊκή εκπαίδευση αστυνομικών. Αυτό που λείπει είναι η κοινή ευρωπαϊκή εκπαίδευση των δικαστών που θα οδηγήσει στην επιστοποίηση των δικαστών και των εισαγγελέων και στο προκείμενο πλαίσιο. Αυτό λείπει και θα πρέπει και αυτό να περιληφθεί γιατί είναι σημαντικό οι δικαστές να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και όχι μόνο οι ανακριτές. Οι δικαστές αλλά ιδίω οι δικάζοντες δικαστές, όπως τους ονομάζουμε εμείς στο δικό μας σύστημα. Οι δικαστές οι οποίοι θα δικάσουν την υπόθεση, να αντιληφθούν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα προβλήματα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ενώσεως. Για τον ΕΠΟ, για τον, εισαγγελέα, τον, Ευρω... τον Ευρωεισαγγελέα δηλαδή, είπαν ορισμένοι ότι ακούγεται η γνώμη ότι δεν τον χρειαζόμαστε. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι τον χρειαζόμαστε. Άρχισε ήδη η προσπάθεια αυτή εδώ και 10-15 χρόνια. Τώρα όμως έχει γίνει απαραίτητη και υπάρχει και τώρα ανοιχτό παράθυρο ευκαιρίας να πιστούν και οι εθνικές αρχές. Εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση, νομίζω ότι μπορεί να πετύχει. Εφόσον είναι σωστές οι συνθήκες πλαίσια, οι αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες. Νομίζω εμείς Είμαστε υπέρ και ο συνάδελφός μου εδώ. Αλλά χρειάζεται μπορεί να σκεφτεί κανεί και διάφορε παραλλαγέ. Ένα εθνικό ευρωεισαγγελέα σε συνεργασία με έναν ευρωπαϊκό ευρωεισαγγελέα και ούτω καθεξή. Πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Είπατε πριν ότι σημειώθηκαν δύο υποθέσεις στο Λουξεμβούργο και υπήρξε μια καταδίκη. Δεν είναι και τόσο άσχημο αυτό γιατί αυτό σημαίνει 50% επιτυχία. Το άλλο 50% ωστόσο δεν έμεινε πουθενά στα αρχεία. Βρίσκεται στη φάση της επεξεργασίας. Σίγουρα την επόμενη χρονιά θα γίνει. Τώρα εμείς βεβαίως έχουμε τα τρία θεσμικά όργανα. Πάρει μην, ελπίζω να πάρουμε και την Γενική Εισαγγελία Υπάρχει και ένα έγγραφο ήδη από τη δεκαετία του 60 που ε, λέει κάπου και στις συνθήκες ότι ό,τι είναι δικαστικό όργανο έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο. Τέλο πάντων, εγώ δεν είμαι πολιτικό, αλλά πάντω αυτό που θα πω είναι το εξή. Πολλέ από τι υποθέσει αυτέ είναι διεθνού χαρακτήρα. Άρα υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών με την αλλοδαπή. Δεύτερο, είναι και θέματα ασυλίων. Τα θέματα των ασυλίων είναι πολύ σημαντικά. συνάδελφοί μου οι οποίοι ασχολήθηκαν με υποθέσει και Ευρωπαίων αξιωματούχων που έχεραν ασυλία, υπήρχε το πρόβλημα εκεί. Και για του ευρωβουλευτές το ίδιο. Και είμαι υπερήφανο που μπορώ να πω ότι οι δικοί μα ευρωβουλευτές έχουν παρετηθεί τη κοινοβουλευτική του ασυλία. Μόνο ό,τι έχει σχέση με την αυστηρή άσκηση των πολιτικών του καθηκόντων, διότι ένας μεθυσμένο ευρωβουλευτή που οδηγεί το αυτοκίνητο θα διώκεται οποιο οπωσδήποτε άλλος ε, ε υπήκος χώρα. της χώρας. Ε, θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο. Θα περάσω το λόγο στο συνάδελφό μου, αν επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ζανό θα ήθελα να προσθέσω ότι στο Λουξεμβούργο ισχύει πολύ υψηλό επίπεδο αλκοολημίας 0,5-0,6 κατά την οδήγηση. Α, 0,5. Ε, επιτρέπεται υψηλό ποσοστό είναι το στο αίμα. Στο Λουξεμβούργο τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να δώσω το λόγο στο δεύτερο καλεσμένο μας, στον εκπρόσωπο του Ισπανού Γενικού Εισαγγελέα, στον κύριο Χόρχε Εσπίνα Ράμος. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να δώσω απάντηση στα σχόλια και των δύο βουλευτών που σχετίζονται λίγο πολύ με τα ίδια προβλήματα. Όσον αφορά τη χαμηλή απόδοση, τους μικρούς αριθμούς σε εθνικό επίπεδο το πρώτο που παραδέχτηκα είναι ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα. Αν ήθελα να περιγράψω με κάποιο τρόπο το συνέστημα που στην υπηρεσία μας, στην Ισπανική Υπηρεσία εισαγγελία είναι απογοήτευση. Εργαστήκαμε πολύ, προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τις υποδομές. Και παρόλα αυτά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των υποθέσεων αυτών είναι η διεθνής διάσταση, η υπερεθνική διάσταση που δεν είναι πάντα παρούσα με τις υποθέσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ισπανία. Έχουμε και καθαρά εσωτερικές υποθέσεις. Και αν αυτές ήταν ο κανόνας, τότε Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Υπηρεσία δεν θα χρειαζόταν. Ξέρουμε όμως ότι δεν ισχύει αυτό. Και έχω την εντύπωση καμιά φορά ότι ο κίνδυνος που ανέφερε ο κύριος Κέσλερ να γίνεται πραγματικό φόρουμ shopping από τους ε, διάφορους εγκληματίες ε, ίσως να ισχύει στην περίπτωσή μας. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε όλες τις υποθέσεις πιφ στην Κεντρική Υπηρεσία της Αγγελίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Έχουμε ένα σύστημα που βασίζεται στον δικαστή που ερευνά τις υποθέσεις και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν συζητάμε την κατάσταση που κρατεί συγκεκριμένα στην Ισπανία. Αν ήθελα να σας πω γιατί είναι χαμηλή αποδοτικότητα, δεν μπορώ να σας πω γιατί ακριβώς. Ακριβώς αφού καταβάλαμε χρόνο και προσπάθεια για όλα αυτά, μην έχοντας δει βελτιώσεις και αποτελέσματα, ίσως γι' αυτό αισθανόμαστε ότι χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό ε, που προτείνεται. Η Ευρωπαϊκή εισαγγελική υπηρεσία, αν υπάρχει συγκέντρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν δοθεί υψηλή ιεραρχική σημασία σε αυτόν τον φορέα, ίσω κάτι να γίνει. Παράλληλα προσπαθούμε να βελτιώσουμε τι επιδόσεις. Έχουμε συμπεριλάβει και την Όλαφ για θέμα για κατάρτιση, αρχική και συνεχή κατάρτιση για του αγγελεί. και ίσως αυτό να αποδώσει εν καιρό καρπούς. Βασικό πρόβλημα με το παρόν σύστημα είναι το εξή. Η Όλαφ μπορεί να διεξαγάγει μόνο διοικητικές έρευνες και καμιά φορά οι έρευνες που ξεκινά η Όλαφ είναι ποινική φύσεως ευθύ εξ αρχής. Παρ' όλα αυτά ξεκινά έρευνες η Όλαφ και όταν λαμβάνουμε τα αποτελέσματα δεν είναι μόνο που δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Αν ξέρει κάποιο ότι ελέγχεται, ερευνάται ακόμα και σε επίπεδο διοικητικό, κάποιο ή κάποια, όπω είπε και ο συνάδελφό μου πριν, πολλέ δυνατότητε που θα είχε όσον αφορά την ποινική δίωξη είναι πλέον Δεν έχει ε, δεν έχει νόημα να διατάξει κατοίκων έρευνα αν κάποιο ε, ήδη ξέρει πριν, ότι πριν από έξι μήνε ξεκίνησαν έρευνα από την όλα αυτών. Θα έχει ακόμα και πρόβλημα να πείσει ένα δικαστή να εγκρίνει ένα τέτοιο μέτρο διζητικό, αν είναι σίγουρο ότι δεν ε, θα μπορέσει κανείς να συλλάβει αυτόν τον άνθρωπο και με τα διάφορα έγγραφα που πιθανόν δεν θα υπάρχουν πλέον. Αυτά τα προβλήματα βλέπουμε με το παρόν σύστημα. Από αυτά θα απαλλαχθούμε αν έχουμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Υπηρεσία. Διότι η δικαστική αστυνομία ε, δίωξη οικονομικού εγκλήματο, α την πούμε όπω θέλετε, θα είναι η Όλαφ και θα υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Τώρα σε σχέση με τις εθνικές διώξεις. Δεν θα είναι συμφωνία μεταξύ Ευρωπαίου εισαγγελέα και των εθνικών εισαγγελέων να αποφασίζουν να κάνουν κατά περίπτωση. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να υπάρχει σαφής ιεράρχηση. Ποιο δίνει εντολέ θα πρέπει να είναι καθορισμένο ιεραρχικά. Και μόνο όταν πέφτει κάτι εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα θα πρέπει ο εκπρόσωπος, να, ε, ο εθνικός, να ακολουθεί τις εντολές του Ευρωπαίου Εισαγγελίου και οι εθνικές συγκελικές αρχές δεν θα έχουν λόγο. Είναι θέμα ποιος θα είναι αρμόδιος για την έρευνα και τη δίωξη συγκεκριμένης υπόθεσης, συγκεκριμένου τύπου υποθέσεων. Τριβές ίσως να προκύψουν και πιθανότατα θα προκύψουν. Οπότε, γι' αυτό το μοντέλο που ανεπίσημα προτείναμε εντό αγωγικών ήταν ένα μοντέλο που μιλούσε για την ανάγκη να υπάρχει ένα βήμα κατάλληλο, ώστε οι γενικοί εισαγγελείς οι διευθυντές των αρμόδιων φορέων έχουν άμεση σχέση, επαφή με τον Ευρωπαίο, Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα για να μειώνονται οι τριβές. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και το Συμβουλευτικό Φόρουμ που συνεδριάζει κανονικά κάθε εξάμεινο στην έδρα του Eurojust στη Χάγη, στη Χάγη για να κάνει αυτό το έργο. Υπάρχουν και άλλες πιθανότητες. αλλά δεν θα χρειάζεται συμφωνία κατά περίπτωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Υπηρεσίας και των Εθνικών Εισαγγελικών Υπηρεσιών. Αυτό θα αντέβαινε σε εξουσίες του Ευρωπαίου, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής. Θα ήταν σαν να παρακαλάμε κάθε φορά να γίνονται αποδεκτές οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής. Αν δημιουργηθεί αυτή η αρχή θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει πλήρεις εξουσίες. Όσον αφορά το Eurojust, αναφέρατε κάτι που είναι λίγο δυσεπίλητο. Τι είναι η συνθήκη όταν λέγει α, ότι από την Eurojust, ότι υπάρχει από Eurojust. Γιατί ένα άρθρο που αναφέρεται στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης αναφέρει το Eurojust και όχι την OLAF, Την Ευρωπόλ που είναι υπηρεσία συλλογή πληροφοριών και όχι την Όλαφ. Ο καθένας μπορεί να έχει τη θεωρία του γιατί υπάρχει αυτή η αναφορά. Η μόνη λογική λύση θα ήταν να θεωρήσουμε ότι αυτό που σημαίνει είναι ότι θα πρέπει να βασιστούμε στην εμπειρία που έχει συσσωρεύσει μέχρι τώρα η Eurojust σαν φορέας δικαστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή είναι φορέας δικαστικής συνεργασίας είναι πολύ Σημαντικό φορέα, Αν δεν είχαμε τη Eurojust θα έπρεπε να είχαμε φεύγει αυτό το φορέα. Αφορά τη συνεργασία όμως μεταξύ ισοτήμων. Η Ευρωπαϊκή Δικαστική Υπηρεσία, Ευρωπαϊ... ο Ευρωεισαγγελέα θα είναι κάτι διαφορετικό. Θα έχει τη δυνατότητα να ξεκινά την ποινική δίωξη και να φέρνει κάποιον στη δικαιοσύνη ε, στο δικαστήριο κάποια συγκεκριμένη χώρα. Διαφορετικό το πεδίο που καλύπτεται Εκτός αν έχουμε Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία που θα έχει 28 κάτι μέλη, κάτι απίθανο, τα καθήκοντα, οι λειτουργίες ήταν διαφορετικές και πάντα θα υπάρχει λόγος να παραμείνει το Eurojust για τα κράτη-μέλη εκείνα που θα αποφασίσουν να μην συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή ε, Εισαγγελική Υπηρεσία. Στο άρθρο 85 υπάρχει δυνατότητα να ξεκινούν οι έρευνες πάντα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Και θα ήταν ε, κοινή λογική να βρούμε ένα ρόλο για την όλα, αφού ώστε να χρησιμοποιείται και αυτή στα πλαίσια των νέων εξουσιών που θα θέτει ο νέος κανονισμός, μελλοντικός κανονισμός, θα το αποφασίσουν οι νομοθέτες αυτό. Και αυτό θα είναι ένας τρόπος συντονισμού των δράσεων μεταξύ κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στο EPPO και κρατών μελών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή αυτή Υπηρεσία. Δεν θα είναι πολύ δύσκολο θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα πρέπει να γίνει μια έρευνα σε τρία κράτη-μέλη στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Συγγελική Υπηρεσία. Εκείνε ξεκάθαρα τα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να διεξαχθεί και σε άλλα δύο κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Συγγελική Υπηρεσία. Υπάρχουν πολλά πράγματα προ συζήτηση και προ απόφαση, αλλά είναι σημαντικό να είμαστε ανοιχτόμυαλοι όσον αφορά τι δυνατότητε, διότι δυστυχώ και δεν ισχύει αυτό μόνο για την Ισπανία, το παρόν σύστημα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε κύριε Εσπίνα Ράμος. Φτάσαμε στο τέλος της ακρόασής μας. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας τώρα, τον κύριο Γκάιερ, για να κάνει μια ανακεφαλαίωση και να ολοκληρώσουμε. Ähm, πολύ ευχαρίστω, κύριε Πρόεδρε, λέει ο Γκάιερ. Πρώτα, θα ήθελα να σημειώσουμε και κάπως με εξέπληξε αυτό που είπαν οι δύο τελευταίοι παρεμβάντες. Το κοινοβούλιο είναι πολύ γλωσσό. Και ότι κάποιος τους είπε να μιλούν αγγλικά δεν μπορεί να είναι σωστό. ούτε είναι θέμα διερμηνέων, έστω και αν η ορολογία είναι εξειδικευμένη. Στις ακροάσεις ο κάθε ένας πρέπει να μπορεί να μιλεί την μητρική του γλώσσα. Δεύτερο, ρωτήσαμε εμείς εάν ...η οι δήμονες που βρίσκονται εδώ διαπιστώνουν σημαντικά ελλείμματα στα έγγραφα που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ δεν άκουσα τίποτα σχετικό. Δηλαδή δεν άκουσα ας πούμε σημαντικές υποδείξεις σχετικά με ελλείψεις στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα θεωρώ ότι είναι επαρκής οι βάσεις αυτές, που βεβαίως θα επεξεργαστούμε με λεπτομέρεια. Ο Πέτερ Στρουκ, παλαιός κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος στην Bundestag, είχε πει ότι τίποτα δεν βγαίνει από το κοινοβούλιο όπως μπήκε. Το ίδιο ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα εξετάσουμε λοιπόν, πολύ προσεκτικά το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάτω από το φως των όσων ακούσαμε. Από την όλα άκουσα ότι θέλουν παραπάνω προσωπικό και λιγότερες εκθέσεις. Το λέω έτσι λίγο οξυμένα. Εγώ θα ήθελα βέβαια να ακούσω μερικές συγκεκριμένες υποδείξεις από την Όλαφ, όπως άκουσα τώρα από τους κύριους Νίσης και Ράμος. Πού βλέπει η Όλαφ να εντοπίζονται τα προβλήματα στη συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Πού πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Πού πρέπει ενδεχομένως να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία να ενισχύσει τα όργανα αυτά. Ενώ δηλαδή τους εισαγγελείς. Εάν τώρα οι εθνικές αρχές, οι εθνικές εισαγγελικές αρχές μπορούν να συνεργαστούν με μια κοινή ευρωπαϊκή, τότε κοινέ προδιαγραφές εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα, όπως είπαν οι εθνικοί εισαγγελείς, ότι οι εισαγγελίε δηλαδή δεν διατηρούν επιφυλάξεις απέναντι στον ενδεχόμενο, στον ενδεχόμενο θεσμό του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα, του Ευρωπαίου συγγνώμη, Εισαγγελέα. Το ερώτημα είναι βέβαια στη βάση ποιων προτύπων θα γίνει η συνεργασία αυτή, ποιον στάνταρτ, καθώς επίσης τίθεται και το θέμα της γλώσσας. Εάν θέλουμε βέβαια να εξετάσουμε την προσέγγιση των εθνικών εισαγγελικών αρχών στις υποθέσεις, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τις προσεγγίσεις αυτές. Και φοβούμαι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο παρά μόνο με υποβολή εκθέσεων. Αλλά ελπίζω να μην τις κάνει όλα αυτές. Από την διεθνή διαφάνεια άκουσα ότι εξακολουθεί να υπάρχει διαφάνεια, ε, συγγνώμη, με εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στις δαπάνες. Δεν περιμένω να ακούσω τίποτε άλλο βέβαια από την διεθνή διαφάνεια παρά να ζητεί περισσότερη διαφάνεια. Σωστό. Συγκρίσιμες εκθέσεις για υποθέσεις απατών επίσης μου φαίνεται πολύ σωστό. Άκουσα πολλά σχετικά με το τι πρέπει να προσέξουμε στη συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Για παράδειγμα, παραπέρα κατάρτιση ε, εθνικών εισαγγελίων και δικαστών σε θέματα δικονομικά αλλά και δικαιοδοσιών. Πιστεύω ότι στο τέλος της προσπάθειας αυτής μπορεί να προκύψει ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και των απατών. Αναμείνω λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον και χαρά την συνεργασία και ευχαριστώ όλες και όλους τους παρισταμένους για τις παρεμβάσεις των. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκάιερ πολύ εύστοχη η ανακεφαλαίωση. Αλλά μία διόρθωση από τη γραμματεία. Δεν επέβαλε γραμματεία ε, της Επιτροπής στα αγγλικά ε, στην συνεδρίαση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Ραντεβού στην επόμενη μας συνεδρίαση.